Καθίστε και παρακαλώ να είστε ήσυχοι, ώστε να μπορέσουμε με ησυχία να προχωρήσουμε. Έχουμε ψηφοφορίες που πρέπει να διεξαχθούν. And the vote will be taking place in this Η ψηφοφορία θα γίνει στην κοινή συνεδρίασή μας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Γυναικών και ΛΥΜΠΕ Πολιτικών Ελευθεριών για την έγκριση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Θυμάτων εγκλημάτων. Γνωρίζετε ότι μετά από μακρότατες και σε βάθος έντονες διαπραγματεύσεις, οι εισηγητές μας τελικά συμφώνησαν με το Συμβούλιο για κανόνες και κανονισμούς καινούριου για ελάχιστα πρότυπα και υποστήριξη όσον αφορά τα δικαιώματα και την υποστήριξη θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Χάρη σε αυτή την οδηγία λοιπόν όλα τα θύματα που έχουν υποστεί τις επιπτώσεις κάποιου εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποφεληθούν από τις ίδιες ελάχιστες διεργασίες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους με ένα βελτιωμένο επίπεδο αρρωγής, συνδρομής και προστασίας. Θέλουμε να χαιρετήσουμε λοιπόν την ολοκλήρωση αυτών των διαπραγματεύσεων και τη στεναρή δέσμευση από τους εισήγητες χάρη και στις προσπάθειες και των δύο αυτών εισηγητριών εισηγητών και των σκιωδών εισηγητών και εισηγητριών με εξαιρετική δουλειά πετύχαμε. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον πρόεδρο κύριο Γκούσταυσον της Επιτροπής Γυναικών. Θα ήθελε να προσθέσει κάποια σχόλια προτού συνεχίσουμε και περάσουμε στην ψηφοφορία έχοντας ακούσει και τους εισηγητές. Κύριε Γκούσταυσον παρακαλώ έχετε τον λόγο και θα συνεχίσω στα σουηδικά. Λοιπόν, παρακαλώ να φορέσετε τα ακουστικά σας για να παρακολουθήσετε την διερμηνία από τα σουηδικά που θα μιλήσω. Πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν κύριε Πρόεδρε, κύριε Φερνάντε Θαβιλάρ, γιατί συμμερίζεστε μαζί μου και είσαστε συμπρόεδρος σε αυτή την κοινή συνεδρίασή μας, εσείς και εμείς στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Είναι μια ικανοποίηση το ότι βρισκόμαστε όλες και όλοι εδώ για να ψηφίσουμε αυτές τις προτάσεις. Όλοι μας ε, πρέπει να εκφράσουμε μεγάλες ευχαριστίες προς, τους, προς τις Έκαναν εξαιρετική δουλειά. Επένδυσαν τεράστιες προσπάθειες και με την υποστήριξη των συνεργατών τους και συνεργατριών τους φυσικά. Επίσης υπήρξε συνεργασία από την Επιτροπή που μας βοήθησε να καταλήξουμε σε αυτήν την συμφωνία. Ευχαριστώ επίσης και το Συμβούλιο για την ελαστικότητά του που θα μας επιτρέψει να ψηφίσουμε προς έγκριση αυτή την ε, πρόταση που μας ικανοποιεί. Επίσης η ικανοποίησή μου πρέπει να εκφραστεί, διότι σε αυτή την έκθεση έχουμε συμπεριλάβει την προοπτική του φίλου με σαφέστατο τρόπο. Προοπτική φίλου σαφής. Είναι πολύ καλό λοιπόν αυτό και θεωρώ ότι είναι πολύ καλό η αναφορά που γίνεται στην ε, βία των ανδρών και της ε, συμπεριφοράς των ανδρών εναντί των γυναικών και την βία εις βάρος των γυναικών μέσω αυτών των πράξεων. Είναι μεγάλη ικανοποίηση για μένα ότι συμπεριλήφθηκε αυτό. Θέλω να ρωτήσω, οι εισηγήτριες θέλουν να παρέμβουν, η κυρία Παρβάνοβα ή η κυρία Χιμένετ. Εσείς θα αποφασίσετε, θέλετε να παρέμβετε ή όχι. Ε, Yes, σας ευχαριστώ κύριε Γκούσταυσον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εσάς κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Επιτροπή, διότι έδωσε φωνή στα θύματα σε σχέση με αυτή την έκθεση που σημειώνεται μεγάλη πρόοδος για τον χώρο ελευθερίας και ασφάλειας στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε και το Συμβούλιο και την Προεδρία της Δανίας για αυτά τα οποία εμείς θεωρούσαμε ότι είναι οι κόκκινες γραμμές και που έγιναν σεβαστές αυτές για τα δικαιώματα που είναι ιερά και απαραβίαστα των θυμάτων και όσον αφορά και την ενημέρωση και την υποστήριξη και την προστασία ιδίω το δικαίωμα προστασίας για να μην υπάρξει δεύτερη θυματοποίηση με την ατομική αυτή συνεισφορά φορά υπέρ των θυμάτων καταφέραμε να λάβουμε υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες Επίσης και τις ειδικέ ανάγκες που έχουν κάποιοι τύποι θυμάτων και συλλογικών θυμάτων, όπως θύματα τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος, θύματα σωματεμπορίας και εμπορίας ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντική και η συμπερίληψη της συνιστώσας της διαφοράς των του φύλου, δηλαδή σε σχέση με τις γυναίκες. Και χάρη στις προσπάθειες ε, των, της γραμματείας ε, και των υπαλλήλων και των βοηθών που συνεισέφεραν πολύ για την επιτυχία αυτής της ε, έκθεση. Ευχαριστώ επίση και την ε, Επιτροπή Γυναικών και την εισηγήτρια από πλευρά τη ε, την κυρία Αντώνια Παρβάνοβα. Ευχαριστούμε και του χειώδεις εισηγητέ για όλε τι παρεμβάσει και συνεισφορέ του. Ολοκληρώνω. Θα ψηφίσουμε μια έκθεση που στου πολίτε ε, δίνει την εντύπωση και τη συνεισφορά να αισθάνονται πιο ασφαλείς όσον αφορά την, τις επιπτώσεις κάποιων εγκλημάτων. Όχι μόνο στις χώρες τους αλλά και συνολικά σε όλη την Ευρώπη. Μπορούμε όλοι να είμαστε υπερήφανες και υπερήφανοι συνεργαστήκαμε υπέρ των θυμάτων, που είναι, εκείνες που εκείνοι που χρειάζονται περισσότερο αυτή τη σύνδρομη. Έχουμε ένα αξιόλογο αποτέλεσμα και ευχαριστώ για αυτό. Thank you very much, Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, λέγει και κυρία Παρβάνοβα, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τερέσα για την εξαιρετική, εξαιρετική αυτή αποτελεσματική εταιρική σχέση και συνεργασία. Να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές και τα μέλη των δύο επιτροπών μας, διότι αποδείχθηκε, καταδείχθηκε μια πολύ επιτυχή συνεργασία. Έχει μεγάλη σπουδαιότητα η σημερινή αυτή η μέρα. Μετά την έγκριση της συνθήκης Λισαβόνας και την έναρξη σε ισχύ της, έχουμε νομοθεσία τώρα που ε, δίνει δυνατότητα προστασίας ατομικά των πολιτών και των θυμάτων όσον αφορά τα εγκλήματα. Είναι η πρώτη φορά που έτσι συνεισφέρει σημαντικά το Ευρωκοινοβούλιο προωθώντας ε, την, αξιολογική, την αξιολόγηση ακριβώς ε, των αναγκών και επιπτώσεων, αποφασίζοντας για συγκεκριμένες ανάγκες και υπηρεσίες που πρέπει να παράσχονται και ειδική κατάρτιση και εκπαίδευση για όλους που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση ακριβώς θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Είμαι υπερήφανη επίσης για το ότι και οι δύο επιτροπές συμφώνησαν σε όλες τις έννοιες και προσεγγίσεις ε, όσον αφορά την βία εις βάρος των γυναικών και την συνιστόσα του φίλου. Θέλω να ευχαριστήσω την Δανέζικη, την Δανική Προεδρία για τις προσπάθειες που έκανε στο Συμβούλιο για να προχωρήσει το θέμα και από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Είναι αξιόλογη η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Είχαμε πραγματικά επαγγελματική υποστήριξη και συμβουλές πραγματογνωμοσύνης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να ευχαριστήσω και δύο γραμματείες και των δύο επιτροπών για όλη την συνδρομή που μας βοήθησαν. Αυτή η οδηγία οπωσδήποτε θα βοηθήσει και θα φέρει μια μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τα θύματα εγκλημάτων. Και θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες, ελπίζω στο μέλλον, να έχουμε μια τέτοια καρποφόρα γόνιμη συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τους τις δεν θέλω να επηρεάσουμε τα μέλη για το πώς θα ψηφίσουν. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι καλό θα ήταν να μην διατρέξουμε μία-μία τις τροπολογίες ξανά. Φυσικά είσαστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε. Είσαστε κύριοι της ψήφου σας. Ε, θα ήθελα καταρχάς με ηλεκτρονική ψηφοφορία να ψηφίσουμε τις συμβιβαστικές τροπολογίες και αν υιοθετηθούν θα περάσουμε στην τελική ψηφοφορία. Πρώτα, στην 539 Ψηφίζουμε την 539. Τη συμβαστική τροπολογία 539. Έναρξη της ψηφοφορίας. Has everybody voted? Σαν όλοι. Όχι. Λείπουν λοιπόν, δύο άτομα. Ένα. Και τώρα υπάρχει ένας παραπάνω. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε, από ό,τι βλέπω. Πολύ ωραία. Πάμε στην τελική ψηφοφορία. Σελίδα 41. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίζουμε παρακαλώ. Ξεκινάμε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετήθηκε. Πραγματικά υιοθετήθηκε. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Στους εισηγητές καλύτερα. Τέλειωσε αυτή η συνεδρίαση. Ευχαριστώ όλους. Καλό καλοκαίρι σε όλους.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 Hello. Please. Thank you all. Ευχαριστώ όλους. Φεύγουν τώρα τα μέλη της Επιτροπής Γυναικών. Πάντα είναι καλή η στενή συνεργασία. Ειδικά οι δύο επιτροπές συνεργάζονται πολύ καλά μαζί, η ΛΥΜΠΕ και η ΦΑΜ, η Επιτροπή Γυναικών και η Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών. Τώρα, τα μέλη της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών θα ψηφίσουν τις επόμενες εκθέσεις, τα επόμενα κείμενα. Μιλάμε για θέματα που είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Θα ξεκινήσουμε το σημείο 15. Μιλάμε για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Η κυρία Νεχέντ είναι η συγγήτρια. Θέλουμε να υιοθετήσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης. Ψηφίζουμε. Τώρα. Και ξεκινάμε. Ας προσπαθήσουμε να διεκπαιρεώσουμε ομαλά αυτή την ψηφοφορία. Συμβιβασμό 1. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβιβασμό 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβιβασμό 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβιβασμό 4. Υπέρ κατά, αποχές, Υιοθετείτε. Συμβιβασμός 5, υπέρ, κατά, αποχές, Υιοθετείτε. Τροπολογία 15, υπέρ, κατά, αποχές, Υιοθετείτε. 16, υπέρ. Ελέγχουμε την 15 εννοείται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά τη 15. Ξεκινάμε την ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίζουν τρεις παραπάνω από το ΕΛΚΑ, βλέπω. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα εσωτερικά σας ΕΛΚΑ. Εντάξει, τώρα είναι εντάξει. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Πρέπει να ξαναψηφίσουμε. Close now. Πολύ ωραία. 30 υπέρ, 23 κατά. Υιοθετείτε. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 18 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβιβασμός 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβιβασμός 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβιβασμός 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβιβασμός 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβιβασμός 10 υπέρ κατά, αποχές, Υιοθετείτε. Συμβασμός 11. Είχε υιοθετηθεί. Ο συμβασμός 10 έχει υιοθετηθεί, έτσι. Συμβασμός 11. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, Υιοθετείτε. Πάμε στην τροπολογία 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Νομίζω ότι μόνο το ΕΛΚ υπέρ. Αλλά αν κάνω λάθος μπορούμε να το ελέγξουμε. Α, και το ECR ψήφισε υπέρ. Όλοι οι υπόλοιποι ψήφισαν κατά, άρα απορρίπτεται. Πάμε στη 46. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο. Συνολικά. Ηλεκτρονικά. Ξεκινάμε τώρα. Πέρας της ψηφοφορίας. 56 ψηφί υπέρ, καμία κατά, δύο αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Χέντε. Μπράβο σας. Πάμε στην τρίτη ψηφοφορία. Στην ε, πρόταση ε, σχετικά με την ε, δυνατότητα πρόσβαση σε δικηγόρο για, στο πλαίσιο κοινικών διαδικασιών ποινικών διαδικασιών ε, της κυρίας Αντωνέσκου. Λοιπόν, ε, προχωρούμε στην ψηφοφορία και ξεκινάμε. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 45. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα πρώτη ε, συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 σε 2 τμήματα Εισαγωγή και α. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερη συμβιβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές ηλεκτρονικός έλεγχος. Γρήγορα όμως. Για την 89 ξεκινάει η ψηφοφορία. Δύο ΕΛΚ ε, ε, επιπλέον. Ένα τώρα. Μείον ένα. Εντάξει. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε τι γίνεται, πώς πάει. Εντάξει. Λίγη ψηφοφορία. 19 εναντίον 35 απερίφθη. 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε ως την συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος για την 99 ξεκινά και πάλι πολύ ελκ τώρα είναι εντάξει και που καταλήξαμε λίγη ψηφοφορία 27 εναντίον 28, δηλαδή απερίφθη, λυπάμαι. 94, όχι, με συγχωρείτε. 28, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 χωριστή ψηφοφορία ε, για την παράγραφο 1 ε, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 χωριστή ψηφοφορία πάλι το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τρίτο τμήμα τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές απερίφθη τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 109 υπέρ κατά αποχές δεν είναι τόσο σαφές. Ηλεκτρονικός έλεγχος στα γρήγορα πάλι. Ελέγχουμε την 109, ξεκινά η ψηφοφορία. Ένας πάλι ΕΛΚ ε, υπερβάλλων. Τώρα είμαστε εντάξει. Πού καταλήγουμε, λίγη ψηφοφορία. 21 υπέρ, 37 κατά, απερίφθη σαφώς. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 119 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 121 υπέρ κατά αποχές απερίφθεται. 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ηλεκτρονικός με συγχωρείτε ε, σηκώστε τα χέρια για την 33 αλλά άρχεται η ψηφοφορία έληξη ψηφοφορία ηλεκτρονικά υποθέτω 41 υπέρ 16 κατά αν είχατε σηκώσει σωστά τα χέρια σας θα ήταν σαφές και χωρίς ηλεκτρονικό έλεγχο Τώρα όμως είναι σαφέστατο. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. 34 υπέρ. Κατέπεσε. Δεν το βλέπω στον κατάλογό μου. Ίσως εγώ έχω μία λανθασμένη παλιά, ένα παλιό κατάλογο. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πολλές από αυτές έχουν ε, καταπέσει. Η 37 νομίζω τώρα είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 είναι ταυτόσημη Η συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 ε, συμβιβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος ηλεκτρονικά για την 14 συμβιβαστική. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Η 26 υπέρ, 30 κατά, απερίφθη, με συγχωρείτε. Εκατόν σαράντα τρία υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 144 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 146 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 148 υπέρ, κατά,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 αποχές ε, απερίφθη Συμβιβαστική 15. Τι έγινε, έχουμε και την 38, την έχουμε ψηφίσει την 38. Τώρα ε, ε, συμβιβαστική 15, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 152, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 170 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 174 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 175 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Κύριε Πρόεδρε. Έχω μια αμφιβολία σε σχέση με αυτό που ψηφίσαμε. Είχαμε ξεχωριστή ψηφοφορία σε ένα θέμα. Ο ε, συμβιβασμός 17 λέει ο πρόεδρος. Συμβιβασμός 17. Θέλω να επαληθεύσουμε, να μου πείτε ποιο ήταν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Είναι σημαντικό. Είχαμε μια ξεχωριστή ψηφοφορία και μου φαίνεται ότι, ότι δεν εκφράστηκε όπως θα έπρεπε το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να ξέρω τι συνέβη, διότι είναι σημαντική αυτή η ψηφοφορία, είναι σημαντική αυτή η τροπολογία για μας. Πρόκειται για το άρθρο 13, το εδάφιο 13, ξεχωριστή ψηφοφορία. Το καταλάβαμε, το καταλάβαμε κυρία λέει ο Πρόεδρος, μάλιστα. Στον κατάλογο ψηφοφορίας που έχω είναι το άρθρο 13, συμβιβασμός 17 ως τροπολογία, συμβιβασμός 18 διορθώνει ο Πρόεδρος. Και έχω και για τα δύο τμήματα αντίστοιχα σε μια παράλληλη ε, τέτοια στήλη επισημαίνεται ότι είναι ξεχωριστή ψηφοφορία και θα το επαναλάβουμε. Θα το επαναλάβουμε λοιπόν για άλλη μια φορά. Γιατί στο κατάλογο που είχα είναι, δημιουργήθηκε σύγχυση όσον αφορά αυτό το θέμα. Όχι μόνο όσον αφορά την αναφορά στον αριθμό αντί 17-18, αλλά και για το συμβιβασμό που καλύπτει ή δεν καλύπτει και τις δύο αυτούς, αυτές παραγράφους. Θα κάνουμε λοιπόν την ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτα θα ψηφίσουμε την παράγραφο σε σχέση με τη συμβαστική τροπολογία 17 και μετά θα πάμε σε δεύτερη ξεχωριστή ψηφοφορία στις παραγράφους 1 και 3. Πρώτα ξεκινάμε με την παράγραφο 2 της συμβαστικής τροπολογίας 17. Ως είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά λοιπόν. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Παράγραφος 2 της συμβαστικής τροπολογίας 17. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚΑ. Ο, συγγνώμη, από τους σοσιαλδημοκράτες. Ένας παρα... Έχουμε έναν παραπάνω από τους σοσιαλδημοκράτες. Να αφαιρεθεί ένας από τη σοσιαλδημοκρατική ομάδα. Τώρα, τώρα τι έχουμε. Να ελέγξουμε λοιπόν. Πέρας ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα 34 υπέρ, 23 εναντίον εγκρίθηκε. Και τώρα το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Συγγνώμη, όσοι είναι υπέρ, χωρίς ηλεκτρονική ψηφοφορία. Κατά, αποχές. Τώρα είναι σαφές το αποτέλεσμα. Εγκρίθηκε πλέον αυτό. Και αυτό μας ξαναοδηγεί πίσω στην 175 τροπολογία. 175 τροπολογία όπως είμαστε. Τι λέτε, 13, 13, άρθρο 13 στην σελίδα μου. Σελίδα 13, άρθρο 13 στον κατάλογο ψηφοφορίας που έχω. Μάλιστα. Λοιπόν, Τροπολογία 175. Όσοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 177. Υπέρ. 176 πρώτα. Λυπάμαι, ζητώ συγγνώμη. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 177 τώρα. Αποσύρθηκε λέτε. Δεν το βλέπω στον καταλογό μου. Παρ' όλα αυτά αποσύρθηκε λέτε. Λυπάμαι, υπάρχει σύγχυση λόγω αυτού του κατάλογου ψηφοφορία και δημιουργούνται προβλήματα. Τέλο πάντων, εντάξει. Συμβιβασμό 18. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίθηκε. Τώρα η τροπολογία 105 σε, σε τμήματα. Όχι. Όχι. Καταπίπτει λοιπόν. Καταπίπτει επειδή εγκρίθηκε το 18, η συμβαστική 18. Πάμε στη 44 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 1. Υπέρ. Τι, τι είπατε. Θέλετε ομού να ψηφίσουμε από κοινού όλες αυτές. Εντάξει, ωραία. 1 ε, έως 7 ε, ομού υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν αυτές. Και τώρα η τροπολογία 9 ξεχωριστά υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 48 υπέρ με προφορική τροποποίηση, προφορικά υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στην τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 21 συμβιβαστική υπέρ. Συμβιβαστική 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε κάτω στην 51 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 52 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 14 αποσύρθηκε 55 τώρα όχι δικό μου σφάλμα ή αγνοήσαμε την 54 και δεν την ψηφίσαμε. Συγγνώμη λέει ο πρόεδρος για την 54. 54 μετά τη συμβιβαστική 21. Πού είναι η 54? Πού βρίσκεται, τι απέγινε. Δεν βρίσκεται στον κατάλογο μας. Πού είναι? Δεν είναι εδώ. Λυπούμε. Λυπούμε. Λόγω του κατάλογου για την ψηφοφορία και πάλι σας ζητώ συγγνώμη. Κάτι πάει στραβά, έχει πάει στραβά. Εν πάση περιπτώσει, μου είπαν ότι έχετε δίκιο. Εξακολουθεί να υφίσταται η 54 και πρέπει να την ψηφίσουμε. Συμφωνείτε λοιπόν, ψηφίζουμε την 54. Εξακολουθεί και υφίσταται υπέρ της 54. Κατά. Αποχές. Αποχές είπαμε. Απορρίφθηκε λοιπόν η 54. Απορρίφθηκε. Και τώρα πάει. Έσβησε αυτή. Καταποντίστηκε. Λυπούμε γι' αυτό δεν υπερψηφίστηκε. Τώρα πάμε, προσέξτε, πάμε στην 14. Προσέξτε τώρα, γιατί υπήρξαν κάποιες, ε, κάποια σύγχυση λόγω του καταλόγου. Πάμε στην τροπολογία 14, πρέπει να επικεντρωθούμε καλύτερα. 14, ένα τμήμα έχει αποσυρθεί, ένα άλλο εξακολουθεί και υφίσταται και πρέπει να ψηφιστεί. Υφίσταται λοιπόν. Αυτό που υφίσταται και πρέπει να ψηφιστεί, αυτό ψηφίζουμε τώρα. Από την 14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 55 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 56 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 57 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 59 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 60 υπέρ κατά αποχές. Θα ελέγξουμε την 60. Άρχεται ηλεκτρονικά η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 60. Άρχεται. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Τώρα εντάξει τα μέλη του ΕΛΚ. Τι γίνεται, για να δούμε. Αποτέλεσμα 29 υπέρ, 28 εναντίον. Λυπούμε, αλλά εγκρίθηκε, κύριε Μπουσούτιλ, η τροπολογία σας, μάλιστα. Θλιβόμαστε για το ότι εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 61 υπέρ. κατά αποχές. Νομίζω απορρίφθηκε θα έλεγα. Όχι. Εντάξει, ας ελέγξουμε και πάλι. Σηκώνετε τα χέρια σας γιατί ήταν ασαφές το αποτέλεσμα. Ελέγχουμε, ψηφίζουμε την 61 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα πέρας είπαμε. Αποτέλεσμα 30 υπέρ 27 εναντίον. Εγκρίθηκε. Λοιπόν, συμβιβαστική 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 64 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 65 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 66 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 67 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 68 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 69 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 69. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. 69. Τροπολογία. Πέρας ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα 30 εναντίον 26 υπέρ. Απορρίφθηκε. Δεν βλέπω να έχουν σηκωθεί, να έχετε σηκώσει τα χέρια σας αρκετοί. Κουράζεστε, το κατανοώ και αυτό δημιουργεί πρόβλημα, καταδεικνύεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τώρα τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 24 υπέρ λέτε για την 70 απορρίφθηκε μάλιστα Τώρα συμβιβαστική 24. Η 70 εγκρίθηκε, λυπούμε. Η 17 εγκρίθηκε, η 70 απορρίφθηκε. Η 17 εγκρίθηκε, η 70 απορρίφθηκε. 17, εντάξει, εγκρίθηκε. Η 70 απορρίφθηκε. Μάλιστα, εντάξει έτσι. Τώρα, συμβιβασμός 24, εντάξει, υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε θα έλεγα. Εγώ έτσι το είδα. Άρα σε ελέγξουμε. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 24 συμβαστική τροπολογία. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 29 εναντίον 25 υπέρ. Απορρίφθηκε. Και έτσι πάμε τώρα στη συνέχεια στην τροπολογία. Όχι 71, λάθος. Εντάξει, ωραία. Στην 71, 71 λοιπόν, υπέρ. 71, κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 81, υπέρ. Κατά. Α, ίδια πλειοψηφία πάλι, απορρίφθηκε. 20, υπέρ. Όχι, η 72 πρώτα λέγεται στον πρόεδρο. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος 72 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 75 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 76 υπέρ κατά αποχές νομίζω εγκρίθηκε έτσι 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 78 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβιβασμός 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τοπολογία 80 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Πάμε τώρα στην 82 υπέρ κατά αποχές 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και πάμε τέλος τι έχουμε οριζόντια εγκάρσια τροπολογία οριζόντια τροπολογία τι λέει εδώ εντάξει Συμφωνείτε. Όχι κάθετη λοιπόν, έτσι. Οριζόντια. Μάλιστα. Ας ψηφίσουμε οριζόντια. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Και τώρα η τελική ψηφοφορία για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Τελική ψηφοφορία άρχεται ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα 51 υπέρ 2 εναντίον. Τέσσερις αποχές. Μάλιστα. Συγχαρητήρια λοιπόν εισηγητά. Συγχαρητήρια. Και τώρα περνάμε μου έδωσαν έναν άλλο κατάλογο ψηφοφορίας που θα με βοηθήσει, ελπίζω, να αποφύγουμε κάποιες, κάποιες συγχύσεις και προβλήματα ή λάθη. Ψηφίζουμε τώρα. Την έκθεση Τριανταφυλλίδη, λοιπόν. Τι λέτε, όχι. Αλήθεια λέτε. Έκθεση Τριανταφυλλίδη. Α, μάλιστα. Ζητώ συγγνώμη. Έχετε δίκιο. Σωστό, σωστό, ναι. Το σχέδιο έκθεσης για την παράνομη κράτηση ατόμων από τις CIA σε ευρωπαϊκές χώρες συνέχεια που δόθηκε σε έκθεση προσωρινής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συγγήτρια είναι η κυρία Ελέν Φλότρο. Θα ψηφίσουμε τώρα συμβιβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Άφετ 1, όχι, συμβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε παραπέρα. Συνεχίζουμε στην 67 τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 60. Να ελέγξουμε λέτε. Εντάξει. Ελέγχουμε και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 67. 67. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. 25 υπέρ 27 εναντίον απορρίφθηκε. Είχατε δίκιο τελικά. Απορρίφθηκε. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει. Τροπολογία 68 και 69 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ αυτών. Εναντίον. Αποχές απορρίφθηκαν. Θέλετε να ελέγξουμε λέτε. Ας ελέγξουμε λοιπόν. Ψηφίζουμε την 68 και 69 αυτές τις δύο τροπολογίες. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ όμως. Τι έχουμε τώρα, τι γίνεται. Λοιπόν, ένας να αφαιρεθεί από το ΕΛΚ, έτσι. Και τι αποτέλεσμα έχουμε. 29 εναντίον 26 εγκρίθηκαν. Οι 68 και 69. Πάμε στην 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Σηκώνετε τα χέρια όμως παρακαλώ, αλλιώς δεν υπάρχει τρόπος να δει και να κρίνει κανείς το αποτέλεσμα. 74 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 75 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Και πάμε κάτω στον συμβιβασμό 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και πάμε παρακάτω μέχρι το συμβιβασμό 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συνεχίζουμε με τον συμβιβασμό όχι με την τροπολογία 93 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Να ελέγξουμε λέτε. Ελέγχουμε και ψηφίζουμε την 93. 93. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Από το ΕΛΚΑ υπάρχουν παραπάνω που συμμετέχουν. Τώρα 29 εναντίον 26 υπέρ απορρίφθηκε. 94 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Να ελέγξουμε λέτε. Να σηκώνετε τα χέρια παρακαλώ. Από ό,τι είδα απορρίφθηκε με τα χέρια που είχατε σηκώσει. Ελέγχουμε τώρα ηλεκτρονικά, έστω εν πάση περιπτώσει. 94. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ένας από το ΕΚ παραπάνω πάλι. Εντάξει τώρα. Αφαιρείται ένας και τι έχουμε. 29 υπέρ 27 εναντίον. Μάλιστα εγκρίθηκε, αλλά να σηκώνετε τα χέρια παρακαλώ, θα βοηθούσε αυτό. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στην τροπολογία, όχι, στο συμβασμό 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Κατεβαίνουμε και προχωρούμε στο συμβασμό 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην 108 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 109 τοπολογία. Θέλετε να ελέγξουμε την 108. 108, εντάξει, αυτή θέλετε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την 108. 108. Ένας από το εκ παραπάνω ο συνήθως. Τώρα εντάξει είμαστε. 29 υπέρ 26 εναντίον. Εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε μάλιστα. Παρακαλώ όμως να σηκώνετε τα χέρια, εντάξει. Η 110 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 111 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 9. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Κατεβαίνουμε και προχωρούμε στην 116 τροπολογία. 116 εντάξει. Όχι, 113. Ο, καταπίπτει 113 σύμφωνα με τον δικό μου κατάλογο. Καταπίπτει, καταπίπτει. 116 λοιπόν, υπέρ. Κατά, άποχες, νομίζω απορρίφθηκε. Ας ελέγξουμε καλύτερα. Ελέγχουμε, γιατί με τα χέρια δεν ήταν σαφές. 116. Άρχεται η ψηφοφορία. 116. Εντάξει είμαστε. 28-28. Ισοψηφία. Απορρίφθηκε λοιπόν. Μάλιστα. Τροπολογία 119. Πώς είπατε εσείς, συγγνώμη. Τι λέτε. Χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται η παρέμβαση. Αλήθεια. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ, πάλι. Εντάξει, έστω, τέλος πάντων. Αν είναι 29 έναντι 28, 29 υπέρ, τότε εγκρίνεται. Τι να κάνουμε. Είσαστε εναντίον εσείς. Να ελέγξουμε ξανά, να ελέγξουμε. Εντάξει, ψηφίζουμε ξανά την 116. Άρχεται η ψηφοφορία. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία για να είναι εντάξει τα πράγματα. Άρχεται η ψηφοφορία 116. Δύο παραπάνω από το ΕΛΚ. Ένας από το ΕΛΚ παραπάνω. Μα τι γίνεται. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Πάλι ισοψηφία. 28-28. Δεν διορθώνεται, απορρίπτεται. Λυπούμε πολύ. Χωρίς μικρόφωνο η παρέμβαση, δεν ακούγεται. Πρόεδρος. Ουσιαστικά, εσείς είσαστε του ΕΛΚ, έτσι. Εσείς κυρία Βίξτρον, προφανώς πρόεδρε, υπάρχει ένας φτωχός διάβολος που ξέχασε την κάρτα του, την έχει χάσει και ψηφίζει και ξανά ναι, φυσικά και το σημείωσα αυτό, το παρατήρησα. Τι, συμπεριλαμβάνεται δηλαδή αυτή η ψήφος. Μία ερώτηση απλή. Τι κάνουν οι σύμβολοι του ΕΛΚ, θα έπρεπε να μετρήσουν τα μέλη τους για να δουν πόσα είναι παρόντα και πόσα ψηφίζουν. Πρόεδρος, εν πάση περιπτώσει Έχουμε την τροπολογία 116. Αποσύρθηκε αυτή. Συμφωνούμε σε αυτό τουλάχιστον. Περνάμε στην 119 τώρα. Τροπολογία 119. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 10. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε κάτω στην τροπολογία 121. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τι λέτε εσείς, 122, 122 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Να ελέγξουμε την 122, ελέγχουμε την 122, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ένας από το ΕΚ παραπάνω πάλι. Λοιπόν, τώρα εντάξει. Εντάξει, πέρας ψηφοφορίας λοιπόν τώρα, πέρας. Αποτέλεσμα 24 υπέρ 30 εναντίον απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε. Και πάμε στον συμβασμό 11. Όχι, 123 λέτε. Ωραία. Τροπολογία 123. Συγγνώμη λοιπόν. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τι λέτε. 123 είπαμε. Εγκρίθηκε. Να ελέγξουμε τώρα. Ελέγχουμε την 123. Ψηφίζουμε και άρχεται. 123. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. 28 υπέρ, 24 εναντίον. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 11 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 125 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Πάμε τώρα στην 128 υπέρ. Είναι ταυτόσιμες λέγεται. 125 και 126 λέτε. Ταυτόσιμες. Ταυτόσιμες λέγεται στον πρόεδρο. Έχουμε και την 124 ταυτόσιμες όλες αυτές, καταπίπτουν αυτές επειδή η προηγούμενη υπερψηφίστηκε. Ψηφίστηκε. Πάμε στην 128 υπέρ, κατά. Λοιπόν, προσέξτε, να έχουμε το πρόβλημα με τα χέρια, εντάξει που σηκώνεται. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να το αντιμετωπίσουμε. Εν πάση περιπτώσει, Ψηφίζουμε την 128 ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. 128. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Και αποτέλεσμα 27 υπέρ 28 εναντίον. Μάλιστα, απορρίφθηκε. Τώρα τι έχουμε. Την 129 και την 130. Είναι ταυτόσιμες οι δύο αυτές. Υπέρ αυτών λοιπόν. Κατά αποχές απορρίφθηκαν. Να ελέγξουμε. Ωραία, να ελέγξουμε. Ωραία. Ψηφίζουμε αυτές τις δύο ταυτόσημες, 129 και 130. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Και αποτέλεσμα 27 εναντίον, 29 υπέρ. 29 υπέρ, 27 εναντίον. Εγκρίθηκαν λοιπόν. Εγκρίθηκαν. Και τώρα η 134 υπέρ. Κατά. Τι κάνουν οι σοσιαλιστές παρακαλώ. Δεν είδα χέρια να σηκώνονται. Δεν είδα κάποια χέρια. Αν δεν σηκώνεται η χέρια δεν υπάρχει τρόπος να κρίνει κανείς ποιο είναι το αποτέλεσμα ψηφοφορίας. Άλμπρεχτ μπορούμε να ψηφίζουμε μόνο ηλεκτρονικά για να λύνεται το πρόβλημα. Ελέγχουμε τα πάντα ούτως ή άλλως και καθυστερούμε. Λοιπόν, να ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, συμφωνείτε όλοι. Αλλά να σηκώνετε χέρια αν δεν ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ξέρω, κουράζεστε και εγώ κουράζομαι. Αλλά να σηκώνετε τα χέρια. Διαφορετικά δεν μπορεί κανεί να κρίνει αποτέλεσμα ψηφοφορία από το Προεδρείο. Θα σηκώνετε λοιπόν τα χέρια, εντάξει, όταν χρειάζεται. Ωραία. Η 134 λοιπόν, υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε, μάλιστα, 134 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται, 134. Ένας από το παραπάνω, να αφαιρεθεί ηλεκτρονικά. Και τώρα που φτάνουμε, Λοιπόν, να αφαιρεθεί ένας από το ΕΚ που ήταν παραπάνω, να φτάσουμε στα ίσα. Λοιπόν, εντάξει, ένας από το ΕΚ να μην συμμετέχει, να αφαιρεθεί. Παρακαλώ, προσέξτε, εντάξει. Είχαμε έναν από το ΕΚ παραπάνω, πρέπει να αποχωρήσει. Τώρα εντάξει, εντάξει. 29 υπέρ 27 εναντίον εγκρίθηκε. Πρόεδρε, διαδικαστικό αν επιτρέπετε. Θέλουμε να γνωρίζουμε τα μέλη που ουσιαστικά είμαστε παρόντα, ώστε εκείνοι που δεν παρίστανται στην ψηφοφορία να φύγουν από την αίθουσα. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά να γίνεται αυτό, να μας μπερδεύουν και να μας ζημιώνουν κάθε φορά, μας βάζουν τρικλοποδιά. Δεν γίνεται. 135. 135 τροπολογία υπέρ.

εγκρίθηκε 138 και 139 ταυτόσημες υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν όχι, συγγνώμη να ελέγξουμε ελέγχουμε λοιπόν 138-139 ελέγχουμε, άρχεται Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 25 υπέρ, 27 εναντίον απορρίφθηκαν. Πολύ καλά. Τώρα, η τροπολογία 140 και 141 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ αυτών. Κατά αποχές απορρίφθηκαν. Προχωρούμε στην 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην 143 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 143. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά και ελέγχουμε. Ψηφίζουμε την 143. Πέρας ψηφοφορίας. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ πάλι. Ε, παρακαλώ να φύγει ένας από το ΕΛΚ. Τώρα εντάξει, μάλιστα. Ωραία. Πολύ καλά, εντάξει. Λοιπόν, ηλεκτρονικά θα ψηφίζουμε, ψηφίζουμε 29 υπέρ 27 εναντίον εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αιτιολογικές σκέψεις, ε, πρώτη τροπολογία υπέρ, τροπολογία 1, ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 2, άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 3. Άρχεται. Πέρας. Και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Τροπολογία 4. Άρχεται. Πέρας. εγκρίθηκε. Τροπολογία 5. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 6. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 7 και 8 είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Απορρίφθηκαν. Συμβασμός 12. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Και το αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Τώρα η τροπολογία 9. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Τροπολογία τώρα 11. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 13. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. 14 ε, με προφορική τροποποίηση άρχεται. Πέρας ψηφοφορία τώρα. Και το αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 15 τροπολογία άρχεται. Πέρας. και ε, το αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Η 16 άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα ισοψηφία απορρίφθηκε. Η 17 άρχεται. Τι είπατε. Χωρίς μικρόφωνο η παρέμβαση. Δεν έχετε κάρτα εσείς. Τι γίνεται. Καταψηφίσατε υπερψηφίσατε. Ε, τότε εγκρίθηκε λοιπόν. Δεν είναι ισοψηφία. Εγκρίθηκε. Σωστό. Τι λέτε. Παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο στον πρόεδρο. Δεν άκουσαν οι διερμηνείς. Εντάξει. Θα σημειωθεί στα πρακτικά της συνεδρίασης ότι συνέβη αυτό σε σχέση με την ψήφο σας δεν αλλάζει η ψηφοφορία όμως το αποτέλεσμά της. Διαμαρτυρίες από την αίθουσα δεν ακούγονται οι παρεμβάσεις. Δεν ακούγεται. Πρέπει να προσμετρηθεί λέγεται. Δεν ακούγεται η παρέμβαση όμως. Πρόεδρος. Λοιπόν, να επαναλάβουμε την ψηφοφορία, σε αυτό θα συμφωνούσατε. Λοιπόν, ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την ψηφοφορία πάλι. Και έτσι θα προσμετρηθεί, δεν έχετε την κάρτα σας, θα μετρηθεί λοιπόν, προσμετράτε έτσι, θα έχουμε, έχουμε πάλι την ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την τροπολογία 16, ηλεκτρονικά την 16, άρχεται. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας τώρα. Και πράγματι 29 υπέρ, 28 εναντίον. Και έτσι η δική σας ψήφος υπέρ έδωσε το θετικό αποτέλεσμα. Και εσείς άλλος ένας, 30. Εντάξει, δεν αλλάζει το αποτέλεσμα, υπερψηφίστηκε. Η 17 τώρα, άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τώρα η 18 άρχεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 18. Πέρας ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Πάμε στη 19. Άρχεται. Σε, σε δύο τμήματα όμως. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα πρώτα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τώρα πέρας ψηφοφορίας. Πέρας είπαμε και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Πάμε στην 20. Ψηφίζουμε. Άρχεται. Συγγνώμη, το δεύτερο τμήμα βέβαια της 19. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεύτερο τμήμα της 19. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα Απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε λοιπόν. Σωστό. Απορρίφθηκε. Εσείς πώς ψηφίσατε κύριε Ιουτσέκ. Τι λέτε, πώς ψηφίσατε. Υπερψηφίσατε, αλλά παρόλα αυτά πάλι απορρίπτεται με το αποτέλεσμα. Λόγω ισοψηφίας. Τι έγινε με εσά, Τι απέγινε με εσά. Δεν μπορείτε να ψηφίσετε, τι συμβαίνει. Κάνατε σφάλμα. Α, εντάξει. Υπερψηφίσατε όμως, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει πλειοψηφία υπέρ. Εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει η μία ψήφος και η άλλη. Λοιπόν, εγκρίθηκε. Τι λέτε. 30 εναντίον 29. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν αλλάζει. Αν κάποιος κάνει λάθος πρόεδρε δεν πρέπει να έχει αποτέλεσμα στο αποτέλεσμα που βλέπουμε στις οθόνες. Αυτός είναι ένας απλός κανονικός κανόνας διαδικαστικός. Μπορεί να διορθωθεί η ψηφοφορία, αλλά το αποτέλεσμα της προηγούμενης ψηφοφορίας δεν αλλάζει. Αυτό κάνουμε σε τακτά διαστήματα, τακτικά, στην Ολομέλεια. Πρόεδρος, ναι, αλλά... Κυρία Λάτφορντ, εσείς δεν είναι ονομαστική η κλίση, έτσι, με ονομαστική κλίση ψηφοφορία. Καθώς δεν είναι με ονομαστική κλίση ψηφοφορία, η κανονική διαδικασία σηκώνουμε τα χέρια. Και μετράει η γραμματεία πώς είναι υπέρ, πώς είναι εναντίον. Τώρα όταν χρησιμοποιούμε τις κάρτες και ψηφίζουμε με υποκατάσταση της κανονικής διαδικασίας, ε, τότε λοιπόν μετράμε με τις κάρτες. Διαφορετικά θα εμείνω και θα επιμείνω να μετράτε απλώς τα χέρια που σηκώνονται και αυτά να προσμετρώνται μόνο. Σίγουρα θα παρατηρήσατε και θα είδατε ότι ψηφίζαμε πάνω από μια ώρα με τα χέρια και κάποιοι ζήτησαν και ήταν λογικό να έχουμε ηλεκτρονικούς ελέγχους σε διαρκή βάση ή αν κάποιος κάνει ένα λάθος. Εν πάση περιπτώσει λέει η κυρία Λάτφορντ, αλλά λαρφον αλλα διαφορετικα δεν είναι τώρα εδώ με ονομαστική κλίση. Διαφορετικά μετράμε και ξαναμετράμε και Εν πάση περιπτώσει υπάρχει πάντα κάποιο περιθώριο ελαστικότητα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Δεν μπορεί κανείς να είναι τόσο μικρόψυχος και μικρόνους σε κανονισμούς, κανόνες που δεν υφίστανται. Θα συμφωνούσατε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία ώστε να επανορθωθεί το σφάλμα, να διορθώσουμε τα κακό κείμενα. Πρόεδρε, πρόεδρε, το ΕΛΚ είχε, το ΕΛΚ είχε δύο παραπάνω ε, στο 29-30 και έγινε λάθος σε σχέση με μία ψήφο. Ζητήσαμε να υπάρξει διακριτική ευχέρεια από πλευρά σας κάποια κατανόηση. Δεν είπαμε τίποτα για τις 29 όταν υπήρχαν παραπάνω ε, που συμμετείχαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Ας επαναλάβουμε λοιπόν την ψηφοφορία τώρα. Στο δεύτερο τμήμα της τροπολογίας, τροπολογίας 19. Επαναλαμβάνουμε ηλεκτρονικά στο δεύτερο τμήμα την ψηφοφορία. Άρχεται ηλεκτρονικά η ψηφοφορία. Δεύτερο τμήμα της 19. Τώρα πέρας ψηφοφορίας όμως. Ψηφίσατε όλοι, όλα εντάξει, πέρας ψηφοφορίας λοιπόν. Τι βλέπουμε ως αποτέλεσμα, 30 υπέρ 27 εναντίον. Εγκρίθηκε λοιπόν. Και δεν προσμετρήσαμε τον κύριο Ήλτσεφ που σήκωσε το χέρι και ψήφισε υπέρ, αλλά δεν είχε κάρτα. Λοιπόν εντάξει, εν πάση περιπτώσει, 20 τροπολογία, άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 29 υπέρ 28 εναντίον εγκρίθηκε. 21 τροπολογία. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Και αποτέλεσμα 28 υπέρ 29 εναντίον απορρίφθηκε. Πάμε στην το 22 τροπολογία. Άρχεται. Τώρα τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα 26 υπέρ 30 εναντίον απορρίφθηκε. Τώρα η τροπολογία 24 άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. και αποτέλεσμα απορρίφθηκε. 25 τροπολογία. 25. 26, 26 μάλιστα. 26, άρχεται. Πέρας. Και αποτέλεσμα απορρίφθηκε. 27 Άρχεται. 27. Δεν καταπίπτει, δεν κατέπεσε λέει ο πρόεδρος 27. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Και αποτέλεσμα απορρίφθηκε. 28 τροπολογία. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας Αποτέλεσμα. Απορρίφθηκε. 29 τροπολογία. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. Απορρίφθηκε. 30. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 31. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα. Απορρίφθηκε. 32. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας τώρα και αποτέλεσμα απορρίφθηκε. 33. Άρχεται. 33. 33. Εξακολουθεί και υφίσταται. Πρέπει να ψηφιστεί. Άρχεται. 33. Άρχεται είπαμε. Α, πώς αποσύρθηκε λέτε. Ο συμβασμός αποσύρθηκε. Η συμβαστική τροπολογία, όχι η 33. Ψηφίζουμε την 33 λοιπόν. Τώρα πέρας ψηφοφορίας. Εντάξει. Πέρας ψηφοφορίας στη 33 που ψηφίζαμε. Α, πέρας ψηφοφορίας είπαμε. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. 34. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Κύριε Μισελ, Καταψηφίσατε, τι συνέβη. Υπήρξε κάποιο λάθος. Δεν λειτουργήσε η συσκευή σας, τι συνέβη. Καταψηφίσατε, έτσι. Απορρίφθηκε, εν πάση περιπτώσει, είτε υπεψηφίσατε είτε όχι, εσείς καταψηφίσατε, απορρίφθηκε. Τροπολογία 35, άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 36 με προφορική τροποποίηση. Άρχεται. Μια στιγμή. Άρχεται είπαμε. Τώρα πέρας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 37 άρχεται. 37 ε, είπαμε άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Τώρα είμαστε εντάξει. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 14. Άρχεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 45 τροπολογία. Άρχεται. 45 άρχεται είπαμε. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Αποτέλεσμα. Απορρίφθηκε. 46 άρχεται. Είπαμε άρχεται. 46. Πέρας. Και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 15. Άρχεται. Πέρας. Και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 51 τροπολογία άρχεται σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα της 51 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα τώρα τις 51 άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας τώρα και αποτέλεσμα απορρίφθηκε. 53 άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. Εγκρίθηκε. Και τώρα ψηφίζουμε το κείμενο όπως τελικά τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονικά φυσικά. Άρχεται η ψηφοφορία μας. Τώρα πέρας ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα τελικής καταμέτρησης Ποιο είναι το αποτέλεσμα. 50 υπέρ 2 εναντίον 5 αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Φλότο. Ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα είχαμε τέτοια διαδικασία, αλλά ωραία, τα καταφέρατε συγχαρητήρια. Ήταν δύσκολη η διαδικασία. Ευχαριστούμε για την προσπάθειά σας. Λοιπόν, τώρα δυστυχώς έχω μία υποχρέωση την οποία δεν μπορώ να αποφύγω. Εξού και η κυρία Κίνγκα Γκάλη, συνάδελφος, θα με αντικαταστήσει και θα συνεχίσει με τις ψηφοφορίες. So, the next, uh, Η επόμενη ψηφοφορία, η, κυρία Χολμάγερ. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα απλώς να σας πω ότι στην τροπολογία 5 ε, στον κατάλογο ψηφοφορίας του ΕΛΚΑ υπάρχει ένα μείον ενώ έπρεπε να είναι συν για το ΕΛΚ. Απλούσατε αυτή την υπόδειξη. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε την ε, ε, ψηφοφορία. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά Ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την τροπολογία 11. Ε, δεν έχουν ψηφίσει όλοι. Τώρα λίγοι. 51 κατεψήφισαν. Τροπολογία 13 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ Με συγχωρείτε, λάθος. 29 λέει η πρόεδρος. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παρακαλώ να ξαμψηφίσουμε για 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 ε, υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ μάλλον την 52 θα την ψηφίσουμε αργότερα στη συμβαστική 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά δεν είναι σαφές οπότε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 54 ξεκινάει και πάλι ένας ΕΛΚ πλεονάζων Εντάξει. 29 υπέρ, 24 κατά, 2 αποχές. Οπότε ε, γκρίνεται 55 ε, υπέρ, κατά. Αποχές. Μπορεί να είναι το ίδιο το αποτέλεσμα, αλλά ζητώ και πάλι να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το 55. Λίγοι. 26 υπέρ, 27 κατά, 2 αποχές, απερίφθη. 57 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Μου είπαν ότι έπρεπε να ψηφίσουμε την 56, οπότε πρώτα ψηφίζουμε την 56, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε τη συμβαστική 8, διότι ψηφίσαμε την 7, τώρα είμαστε στην 8, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 69. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. 27 υπέρ, 25 κατά, 2 αποχές, οπότε εγκρίνεται. καταψήφισα και δεν μπορούσα, οπότε τώρα είμαστε 27-27. Γιατί και ο κύριος Λιούτσεφ ήταν κατά, απορρίφθη δηλαδή. 28 υπέρ. Με συγχωρείτε. 68 διορθώνει η πρόεδρος. Υπέρ, κατά, αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 68. Λίγοι. 26 υπέρ, 25 κατά και 2 αποχές. δηλαδή με τον κύριο Ιλτσεφ 26 υπέρ και 26 κατά, οπότε έχει απορριφθεί. Πάμε τώρα στην 73 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται, συμβιβαστική 9 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος ξεκινά για το δεύτερο μέρος της ε, συμβιβαστικής εννέα. Λίγη. 24 υπέρ, 29 κατά, 30 κατά, απερίφθη είστε υπέρ ή κατά, αλλά ό,τι και να είσαστε πάλι απερίφθη. Η κυρία Ντιόν. Με συγχωρείτε. Αλλά νομίζω ότι ξεχάσαμε να ψηφίσουμε μερικές τροπολογίες, διότι το 68 70-71 είχαμε ψηφίσει την 69 αλλά την 70-71-72 νομίζω δεν τις ψηφίσαμε. Λοιπόν, πρέπει να ψηφίσουμε την 70, 71 και 72. Καταρχήν την 70. Ποιος είναι υπέρ. Τροπολογία 70 υπέρ, κατά, αποχές. Είναι πολύ δύσκολο, οπότε ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 70. Λίγη. 25 υπέρ, 28 κατά με μία αποχή. Πάμε στην 71 υπέρ κατά αποχές απερίπτεται και πάλι το ίδιο 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται την 73 την έχουμε ψηφίσει και υπερψηφίσει όπως και τη συμβαστική 9 όπου υπερψηφίστηκε το πρώτο μέρος, καταψηφίστηκε το δεύτερο και τώρα είμαστε στην τροπολογία 75. Εάν λοιπόν συμφωνείτε, παρακαλώ να, είναι, να μου πείτε ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά αποχές είναι δύσκολο. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ξεκινάει. Για την τροπολογία 77. Το ΕΛΚ έχει πάλι έναν πλεονάζοντα. Τώρα είμαστε εντάξει. 25 υπέρ, 26 κατά και 2 εποχές. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απερίφθη. Ας κάνουμε ένα ηλεκτρονικό έλεγχο. Λίγη. 25 υπέρ, 29 κατά. Άρα απερίφθη. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 12. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά πάμε στην 91 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος ξεκινάει Close the vote. 21 in favor, 32 against. I'm sorry. I... Λοιπόν, 92 υπέρ, κατά, Μάλλον 96 ζητά συγγνώμη η πρόεδρος υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Παρακαλώ μπορείτε να ψηφίσετε άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 28 κατά. Απορρίπτεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. πέρας ψηφοφορίας 30 υπέρ, 23 κατά. Μία αποχή εγκρίνεται. 103 υπέρ, κατά. Αποχές υιοθετείται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 111 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι υιοθετείται. Ελέγχουμε την 111. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 41 ψήφι υπέρ, 12 κατά. Καμία αποχή. Συμβιβασμός 15 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 117. Τροπολογία 117 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. Συμβιβασμός. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 17 σε δύο τμήματα. Υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Δεύτερο τμήματα, ε, τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής τροπολογίας 17. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας φοφορίας. 14 υπέρ, 40 κατά. Απορρίπτεται. 118. Όχι λάθος. 122. Διορθώνει πρόεδρος. 122. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 123. Υπέρ. Κατά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ακόμα μια φορά, σηκώστε τα χέρια για την 123 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεν μπορώ να αποφασίσω, το ελέγχω ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 13 κατά, 18 αποχές. Εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 127 υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 127, ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 29 κατά. Απορρίπτεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 129 υπέρ κατά εποχές ελέγχουμε την 129 ψηφίζουμε τώρα πέρας ψηφοφορίας 27 υπέρ 25 κατά υιοθετείται 131 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 132 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά πρέπει να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 36 κατά, απορρίπτεται. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε, 134 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε 135 υπέρ. Κατά. εποχές υιοθετείτε 136 υπέρ. Κατά. εποχές υιοθετείτε 137 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε 138 υπέρ. Κατά. εποχές υιοθετείτε 140 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι υιοθετείτε. Αλλά δεν βλέπω ότι είναι σοσιαλιστική ψήφο. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. 143. Ψηφίσουμε μόνο το δεύτερο τμήμα της 143. Υπέρ. Κατά. Άποχες. υιοθετείτε. 41. Καταπίπτει. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι υιοθετείται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 145. Αρχίζουμε. Τελειώνουμε. 24 υπέρ, 29 κατά. Απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να το ελέγξω ηλεκτρονικά. Συγγνώμη. Αφού δεν σηκώνω τα χέρια, ξεκινάμε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 29 κατά, απορρίπτεται. 147 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 148 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 149 και 150 που είναι ίδιες, υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας, 28 υπέρ, 26 κατά. 27 κατά δηλαδή. Πέρασε πάντως. Τώρα πάμε στη 156 υπέρ. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 159 υπέρ. Κατά. Πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας. 35 υπέρ, 18 κατά. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε τις αντιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρας 25 υπέρ, 29 κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερη τροπολογία υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπέρ. Τρίτη τροπολογία, συγγνώμη, υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. Έξι υπέρ. Κατά. αποχές το ελέγχουμε ηλεκτρονικά, το, την έκτη τροπολογία, τώρα, πέρας 25 υπέρ, 29 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά. Αποχές υιοθετείτε. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Συμβιβασμός 18 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Εγκρίθηκε. Συμβαστική τροπολογία είναι υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Έναρξη. Πέρας. 47 υπέρ. 4 κατά 2 αποχές. Συγχαρητήρια. Τελευταία ψηφοφορία για σήμερα είναι το σχέδιο γνωμοδότησης για τις μόνιμες κυρώσεις για άτομα που κάνουν χειραγώγηση της αγοράς με εισηγήτρια την κυρία Μποσκούρτ. Ψηφίζουμε αμέσως, αν δεν θέλει η κυρία Μποσκούρτ να μιλήσει, με την τροπολογία 17 και 18 που δεν είναι αποδεκτές. Ξεκινάμε με την τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 4 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 5 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 19 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 20 αποσύρεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, διαθετείτε. 8 αποσύρεται, 21 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 23 υπέρ, 8, κατά, αποχές, υιοθετείται. Πάμε τώρα στα εκτιμώντα και τις ιατρικές σκέψεις. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Και τώρα πάμε στην ε, τροπολογία 10 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται, 11 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται, 12 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται, 13 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται, συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται, τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται, 2 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται, συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Και τώρα πάμε στη τελική ψηφοφορία που είναι ηλεκτρονική έναρξη. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. 45 υπέρ. ένα κατά. Τέσσερις αποχές. Συγχαρητήρια και Σκούρτα. Τώρα.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 Θα δώσω το λόγο στον κύριο Φοντάνα τώρα, με συνεχεία στην Κομισιόν και στην Κυπρική Προεδρία για τα σχόλιά της. Κύριε Φοντάνα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κανονισμός επί του οποίου η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ πρέπει να αποφανθεί, θα ισχύσει για το Ταμείο για, την, για το άσυλο και τη μετανάστευση και την εσωτερική ασφάλεια με βάση το χρονοδιάγραμμα 14-20, όπου κάθε Ταμείο έχει τις δικές του γενικές διατάξεις. Η Κομισιόν τώρα προτείνει ένα κανονισμό οριζόντιο που θα ισχύσει σε όλα τα ταμεία. Αυτός ο κανονισμός είναι τμήμα ενός πακέτου τεσσάρων κανονισμών που θα αποτελέσουν το πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εσωτερικές υποθέσεις, ρυθμίζοντας τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, τον έλεγχο και το κλείσιμο των προγραμμάτων καθώς και τον απολογισμό. Όλα αυτά τα στοιχεία δηλαδή. Οι τροπολογίες που είναι γενείς αυτού του κανονισμού που θέλω να προτείνω στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ βασικά ε, κινούνται γύρω από τρεις άξονες. Η έμφαση που δίνεται στην αρχή της επικουρικότητας, την εμπλοκή των τοπικών αρχών στην διαδικαστική φάση, ούτω ώστε να υπάρξει μια μεγαλύτερη απλούστευση της χρήση του δημοσιονομικού, του χρηματοδοτικού μέσου, χωρίς όμως να μην γίνουν οι έλεγχοι που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Οι περισσότερες τροπολογίες που έχουμε παρουσιάσει βάζουν την έμφαση την, στην αρχή της επικουρικότητας. Εκεί που ζητάμε το συγκεκριμένο πλαίσιο κάθε κρατούς μέλους να ληφθεί σοβαρά υπόψη ε, σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Στο άρθρο 3, η πρόταση της Κομισιόν περιοριζόταν σε μια ασθενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Για αυτό το σημείο μας φαίνεται σημαντικό να προσθέσουμε ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι πολίτες να συμμετέχουν. Ε, η αρχή της Επικουρικότητα παίζει ήδη και συνδέεται και με την αρχή της διαφάνειας. Όταν ε, ένα κράτο μέλος θέλει να αυξηθεί η χρηματοδότηση στο 90% είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη αυτές τις αρχές. Επίσης, το ενδιαφέρον κράτο μέλο, θα πρέπει να παρουσιάσει την απαραίτητη τεκμηρίωση και να δικαιολογήσει με λεπτομέρεια το αίτημά του. Άρθρο 16, παράγραφος 4. Επίσης, θέλουμε οι περιφερειακές τοπικές αρχές και οι πολίτες να αποτελέσουν ένα ε, στήριγμα για την Κομισιόν για να βελτιώσει την ποιότητα των ελέγχων, χωρίς να περιοριστούμε στη σχέση απλώς Κομισιόν ε, κατά τους μέλους. Άρθρο 29.5.2. Επίσης, για την υιοθέτηση των ε, διατάξεων για να υπάρξει αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων ελέγχου και διαχείριση. Άρθρο 29, παράγραφος 6. Για αυτό το λόγο, μπήκαν δύο τροπολογίες με τις οποίες ζητάμε η Κομισιόν να αναλάβει, να δημιουργήσει ένα σύστημα παρακολούθησης σε κάθε ταμείο σε ό,τι αφορά την βοήθεια έκτακτης ανάγκης, από τη χορήγηση των πόρων μέχρι την χρήση τους, άρθρο 8, παράγραφος 4, νέα παράγραφος. Και να υπάρχει ο ίδιος μηχανισμός παρακολούθησης σε ό,τι αφορά τις δράσεις για τις τρίτες χώρες, άρθρο 9, παράγραφος 2α νέα. Επίσης παρουσιάστηκαν τροπολογίε για να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στον αποφασιστικό ρόλο ή σε ορισμένε περιπτώσει ενημερωτικό ή συμβουλευτικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φερρυπίν, άρθρο 7, παράγραφο 1. 8, 1, 13, 1, 1. Σε ό,τι αφορά το ρόλο του Κοινοβουλίου, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η εμπλοκή ημών των Ευρωβουλευτών δεν σημαίνει παράταση των προθεσμιών. Όταν η Κομισιόν αποφασίσει να δώσει έκτακτη βοήθεια, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τουλάχιστον εμείς έτσι το έχουμε σκεφτεί, θα πρέπει να ενημερωθούν. Άρθρο 8, παράγραφος 4. Επίσης έχουμε μία σειρά από τροπολογίες για να ενισχύσουμε αυτές τις αρχές για τις οποίες μόλις μίλησα. Επίσης προσπαθήσαμε να μην αλλοιώσουμε το κείμενο της Κομισιόν που μας φαινόταν ούτως ή άλλως καλό για μας. Όμως προσπαθήσαμε να το χτενίσουμε και να εμπλέξουμε τις τοπικές αρχές πέρα από τα εθνικά κράτη. Βεβαίως ξέρουμε ότι τα 27 κράτη-μέλη έχουν διοικήσεις τελείως διαφορετικές και δεν θα είναι για όλους εύκολο να εμπλέξουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Αλλά όμως Εμεί λειτουργήσαμε με την αρχή τη ε, επικουρικότητα. Δηλαδή, κάθε κράτο από εκεί και πέρα μόνο θα δει με ποιο καλύτερο τρόπο θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Εγώ είμαι στη διάθεσή σα για σχόλια και κριτικέ, επικοδομητικέ κριτικέ. Σα ευχαριστώ και σα δίνω το λόγο. Τώρα στρέφομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού ευχαριστήσω τον εισηγητή για τα σχόλιά του θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να αναφερθώ και να απαντήσω σε ορισμένα θέματα τα οποία έθιξε. Χαιρετίζουμε το ότι ε, τόνισε τον ρόλο των αρχών ε, στην εφαρμογή αυτών των ε, ταμείων και στις ε, συνεργασίες μεταξύ κρατών μελών. Οπότε και πάλι θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή παρόλο που ο ρόλος των κρατών μελών για τον έλεγχο δεν πρέπει να μειωθεί την ε, ε, παραπομπή της ευθύνης αυτής σε τοπικές αρχές γι' αυτό και ε, όταν γίνεται αναφορά σε μικρότερες, μικρότερους εκπροσώπους των εθνικών αρχών θα ήθελα να τονιστεί αυτό. Επίσης το άρθρο 13 όπου αναφερόμαστε στον ρόλο ο των εθνικών αρχών όπου προτείνεται να επανεξεταστεί το εθνικό πρόγραμμα. Τα προγράμματα τα οποία έχουν καταρτιστεί μπορούν να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες. Θα θέλαμε να υπάρξουν πολυετή προγράμματα τα οποία δεν χρειάζεται να ανανεώνονται συχνά διότι αυτό θα διαταράξει τις δραστηριότητες και την αρχή των πολυετών προγραμμάτων που είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό των ταμείων αυτών. Θα ήθελα λοιπόν να συνοψίσω τις ε, βασικές ανησυχίες που έχουμε σχετικά με την έκθεση του εισηγητή. Καταρχήν αυτό που είπαμε σήμερα το πρωί για το εσωτερικό ταμείο ασφαλείας και την μεσοπρόθεσμη ε, ε, αναθεώρηση η οποία προτείνεται να γίνει τον Ιούλιο του 2016. Κατά τη γνώμη μας είναι πολύ νωρί διότι τα περισσότερα προγράμματα θα ξεκινήσουν το 2014 και είναι πάρα πολύ δύσκολο τον Ιούλιο του 2016 να αξιολογήσουμε αν χρειάζονται τροποποιήσεις χρηματοδοτήσεως και των προγραμμάτων και θα χρειαστεί να υπάρχουν οι εκθέσεις μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2014 βάσει των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση. Θα ήθελα λοιπόν ο εισηγητής ε, να σκεφτεί αυτή την ημερομηνία, τη λάβει υπόψη και αυτό ισχύει και για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας και την δικιά του μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση. Όσον αφορά την έκτακτη βοήθεια, όπως ε, είπε ε, και το Κοινοβούλιο, όταν χορηγείται έκτακτη βοήθεια σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, θα πρέπει ε, ε, να γίνεται αυτό μετά από ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Δηλαδή δεν θέλουμε μεν να καθυστερήσουμε την ε, χορήγηση έκτακτης βοηθείας αλλά να υπάρχει σωστή ενημέρωση. Όσον αφορά το κάθε ταμείο και το σύστημα χορήγησης βοηθείας εκτάκτου ανάγκης θα πρέπει να υπάρχει μία στενή παρακολουθήση γιατί ε, υπάρχει ένα ειδικό σύστημα εδώ για να παρακολουθείτε αυτή η βοήθεια. Πέραν αυτού θέλω να πω ότι στον πολιτικό διάλογο χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα δώσουν τη δυνατότητα να υπάρξει ένας διάλογος με κάθε κράτος μέλος του χρόνου πριν από την κατάρτιση του προγράμματος για τα δύο ταμεία και ε, μετά από την ανακοίνωση ε, με την οποία θα κοινοποιήσουμε στον, ε, στο Κοινοβούλιο τα πορίσματα του διαλόγου αλλά θα θέλαμε να υπάρξει καταρχήν ο διάλογος και γι' αυτό θα συζητήσουμε με τον εισηγητή για να δούμε πώς θα προχωρήσει η ενημέρωση του Κοινοβουλίου. Όσον αφορά την τροπολογία 15 και 16 και τα εθνικά προγράμματα, ο εισηγητής θέλει να αυξήσει τη λεπτομερή περιγραφή των προγραμμάτων και να υπάρχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με ε, τον λεπτομερή προϋπολογισμό. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι βασικό να έχουμε βασικά στατιστικά στοιχεία, αλλά πρέπει να υπάρχει και μία ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ε, αποφυγή δεσμευτικών προγραμμάτων τα οποία θα έπρεπε να αλλάζουν όλη την ώρα. Αυτή είναι η αρχή την οποία προσπαθούμε να προωθήσουμε βάσει αυτών των προγραμμάτων εξού και παρακαλώ τον εισηγητή να το λάβει υπόψη του. Και όσον αφορά την τροπολογία 23, προτείνει ο εισηγητής να, η ελεγκτική αρχή να είναι μια εθνική, ε, μια ιδιωτική εταιρεία. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι δημόσια για να υπάρχει μία έγκυρη απόφαση ε, όσον αφορά την ε, ε, επιβεβαίωση της ε, ε, σωστής διαχειρίσεως. Βεβαίως ε, αντιλαμβανόμαστε τη σκέψη του εισηγητή αλλά πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν να ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία. Θα σταματήσω εδώ και είμαι στη διάθεση του εισηγητή αν θέλει να συζητήσουμε τις διάφορες τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Φλωρίδης. των τεσσάρων προτάσεων κανονικών. Όπως έχω ήδη αναφέρει, σχετικά με τη διαχείριση των τεσσάρων προτάσεων κανονισμών εσωτερικών υποθέσεων του πολιετούς δημοσιονομικού 1420, η Κυπριακή Προεδρία έχει συστήσει μια κοινή ομάδα για, την, για τους εν λόγω κανονισμούς. Στόχος είναι ο καλύτερος συντονισμό και ειδικότερα των τριών τομεακών κανονισμών σε σχέση με τον οριζόντιο, που θέτει και τις βάσεις για το συνολικό σύστημα διαχείριση των δύο ταμείων. Συγκεκριμένα, αναφορικά με την πρόταση για τον οριζόντιο κανονισμό, το Συμβούλιο έχει ήδη πραγματοποιήσει τρεις αναγνώσεις και η Προεδρία προτίθεται μέχρι το τέλος Ιουλίου να έχει συνάντηση των κρατών μελών στη σχετική ομάδα εργασίας. Η στρατηγική που θα ακολουθήσει η Προεδρία συνίσταται στην επίτευξη σύγκληση των υπόλοιπων σημείων για τα οποία δεν υπάρχει ακόμη κοινή θέση προκειμένου να αποκτήσει άμεσα εξιοδότηση από το Συμβούλιο και να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας συναπόφασης με το Κοινοβούλιο μέσα στο φθινόπωρο. Στόχος του Συμβουλίου και των κρατών μελών είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η ευελιξία των κανονισμών κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων. Τέλος, η Προεδρία χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής και τις εισηγήσεις του κυρίου Φοντάνα και ευελπιστούμε σε μια άμεση και καλή συνεργασία για το εξάμεινο της Προεδρίας μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, εκφράζουμε ονόμα της κυρίας Φαγιών, η οποία δεν μπορεί να είναι εδώ. Τα δικά της λόγια μεταφέρω, λοιπόν. Πριν από όλα και λαμβάνοντα υπόψη την ε, περιπλοκότητα της φύσης ε, του κανονισμού, ε, η κυρία Φαγιών θα ήθελε μια πιο έντονη συνεργασία με τον εισηγητή από την πρώτη ανταλλαγή απόψεων που έγινε στις 20 Μαρτίου του 2012 δεν οργανώθηκε καμία ε, συνεδρίαση των σκιωδών. Και το ίδιο συνέβη και με την συνεδρίαση των συμβούλων. Λυπούμαστε γι' αυτό και θα νομίζουμε ότι αυτό θα επηρεάσει την ποιότητα της έκθεσης που θα παρουσιάσει ο εισηγητής. Παρότι το απευχόμεθα. Υπάρχει πρόβλημα, ναι. Bien que très technique, la πολύ τεχνική πρόταση. Παρ' όλα αυτά η πρόταση κανονισμού είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί δίνει μια δομή για τρία ε, δημοσιονομικά μέσα που είναι πολύ σημαντικά για την ασφάλεια, ελευθερία και κρίμα που δεν λαμβάνουμε υπόψη την πολύ σημαντική αυτή διάσταση. Το σχέδιο έκθεσης δεν, λαμβάνει, δεν υπα... περιλαμβάνει αιτιολογική σκέψη που θα μιλούσε για την ουσία ε, του κειμένου θα μα έδινε όλο το πλαίσιο και θα μα επέτρεπε να κάνουμε μια πιο ενδελεχή συζήτηση για την έκθεση. Κάποιε από τι τροπολογίε που προτείνονται είναι πολύ επιφανειακέ, ειδικά σε ό,τι αφορά την ε, τεχνική φύση του σχεδίου κανονισμού και την προπλοκότητά του. Παρότι ε, κάποια από τα σχόλια τη πρώτη ανταλλαγή απόψεων, ε, απόψεων ε, αντικατοπτρίζονται, αλλά δεν έχουν περιεχόμενο. Αυτό ε, οφείλεται στι συνεδριάσει που δεν έγιναν. Και γι' αυτόν τον τρόπο είναι δύσκολο να κάνω σχόλια στον εισηγητή. Πέρα από το ότι η κυρία Φαγιόν θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ στο θέμα αυτό και θα καταθέσει τροπολογίε ε, που είναι ε, κατάλληλε ε, δεδομένη τη ε, περιπλοκότητα και τεχνική φύση του κειμένου. Καταρχά, οι εμπειρογνώμονε, σε μη κυβερνητικέ οργανώσει κτλ. θα πρέπει να συμμετάσχουν στα πλαίσια αυτή τη εταιρική σκέψη για την προετοιμασία, εφαρμογή και παρακολούθηση των εθνικών προγραμμάτων. Η κυρία Φαγιόν θα ήθελε επίση περισσότερε διευκρινήσει για την διάταξη που προτείνεται ε, για την καταπολέμηση τη απάτη και των άλλων παράνομων δραστηριοτήσεων. Ε, Παραδείγματο χάρη για τι πληροφορίε που μα δίνει η Κομισιόν και το γραφείο, και, και, το γραφείο της Όλαφ. Ε, θα συνεργαστούμε ούτω ώστε να εκπονήσουμε αυτέ τι τροπολογίε. Η κυρία Φαγιόν θα ήθελε περισσότερε διευκρινήσει για το πεδίο εφαρμογή και τη λειτουργία τη κατεπίγουσα βοήθεια. Ένα άλλο σημείο επί του οποίου θα ήθελε περισσότερα συγκεκριμένα μέτρα και περισσότερε πληροφορίε ε, να δοθούν στου ε, πιθανού δικαιούχου. Ούτω ώστε να ενημερώσουμε πολύ καλά του δικαιούχου για το στόχο και τι προτεραιότητε των εθνικών προγραμμάτων. Ευχαριστώ.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 Συγγνώμη, άκουσα το όνομα Κέρκοπ και δεν πρόσεξα ότι αναφερόσαστε σε μένα. Γι' αυτό δεν παρενέβη. Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση ευθύ εξ αρχή. Δεν υπάρχει ούτε μια κοινοβουλευτική επιτροπή που να μην είναι τόσο σαφώ ασαφή στον προγραμματισμό όσο σε σχέση με την κοινοβουλευτική επιτροπή ΤΡΕ. Θα πρέπει να διαβιβαστεί σε σχέση με τη γραμματεία αυτή η παρατήρηση με κάθε τρόπο. Να υπάρξει σχεδιασμό ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε αποτελεσματικά Στι Στις 5 είχα ανηλυμένη υποχρέωση. Στι 5.30 ε, ε, ε, είχα υποχρεώσει αλλού. Δεν μπορεί κανεί με αυτόν τον τρόπο να τηρεί την ημερήσια διάταξη. Όχι μόνο για μένα αλλά και για άλλου. δημιουργούνται πάμπολα προβλήματα. Δεν μπορεί αυτό να είναι αποδεκτό. Και σε άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα αν επιτρέπετε. Επιτρέψτε μου να το πω. Τώρα, για κάποιε παρατηρήσει σε σχέση με την έκθεση που θα ήθελα να κάνω. Θετικά θα ήθελα να αναφέρω ότι από πλευράς Φοντάνα ενισχύεται αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από πλευράς γενικών αρχών όσον αφορά συνεκτικότητα, συμπληρωματικότητα, παραπληρωματικότητα όσον αφορά τα κράτη-μέλη και λαμβάνονται υπόψη αυτές οι ανάγκες τους. Θετικό το βρίσκω επίσης σε σχέση με τις γενικές αρχές το ότι η σχέση κόστους-οφέλους, πώς να το πω, υπό το πρίσμα μιας στοχοθετημένης δράσης με βάση αποτελέσματα, θετικά αποτελέσματα και αηφορία πρέπει να δρούμε. Προβλήματα έχω εκεί όπου υποστηρίζονται κάποια πράγματα όσον αφορά κάποιες αρχές και υπηρεσίες στις αναφερόμενες υπηρεσίες στο άρθρο 23, έχω πρώτα μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλήγουμε πραγματικά σε απλούστευση όταν τρεις υπηρεσίες αναφέρονται παράλληλα. Η πρώτη είναι μια υπηρεσία για την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων. Είναι αρμόδια για αυτά. Δεύτερη αρχή που αφορά διοικητικού ελέγχους που επομίζεται αρμοδιότητα. Το τρίτο είναι μια ελεγκτική αρχή, ελεγκτική υπηρεσία. Το θεωρώ αξιόλογο να δούμε το ότι και η ανεξάρτητη ελεγκτική αρχή είναι ιδιώτες που μπορούν να δράσουν εκτός αυτού του πλαισίου. Μπορεί να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν αυτές οι τρεις υπηρεσίες ή οργανισμοί είναι λογικό να υπάρχουν από κοινού και οι τρεις. Έχω επιφυλάξεις και σε κάποια άλλα σημεία για την έκθεση. Και αυτό που ο εισηγητής Φοντάνα αναφέρεται στο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, όπως λέει και οι τοπικές αρχές, περιφερειακές αρχές και δημοτικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους. Δεν ξέρω τώρα πώς στην πρακτική εφαρμογή όλα αυτά θα μπορούν και θα πρέπει να λειτουργήσουν. Εδώ έχουμε τους πιο διαφορετικούς κανονισμούς για τοπικές αρχές και τοπικές αρχές που μπορούν με διαφορετικό τρόπο να λάβουμε υπόψη ότι έχουν διοργανωθεί. Κάποιες χώρες έχουν κεντρικό σχεδιασμό, άλλες χώρες έχουν ομοσπονδιακό σχεδιασμό και δομή. Όλα αυτά νομίζω δεν μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά, δεν είναι λειτουργικά. Και επιπλέον αν είχαμε παντού τις τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές που θα εμπλέκονται και θα εμπλεκόντουσαν, τότε θα πρέπει και άλλα πράγματα να αλλάξουν. Δηλαδή σε αυτές τις τοπικές περιφερειακές και δημοτικές αρχές και αυτές σύμφωνα με την αρχή της οικονομικής αποτελεσματικότητας να μπορούν να εργάζονται και να έχουν αποδόσεις. Δηλαδή ίδιοι και ίσοι κανόνες και διατάξεις για όλους, για όσους εμπλέκονται στις ίδιες διεργασίες και ε, ε, διαδικασίες. Είναι καλύτερο να δούμε σε σχέση με την πρόταση που θα ακολουθήσουμε τα διακρατικά προγράμματα και η βάση τους και η δομή τους. Εκεί η εταιρική σχέση να προωθείται βέβαια. Εκεί οι, εταιρικοί, περιφερειακές αρχές όμως εντάσσονται στις εθνικές ιδιαιτερότητες και όχι στο συνδυασμό ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κρατών Μελών και περιφερειακών, τοπικών και ε, δημοτικών αρχών. Μου φαίνεται ότι είναι πιο πρακτική και πιο αποτελεσματική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με αυτό το πλαίσιο. Επίσης, και αυτό πιστεύω ότι συμφωνεί με το προηγούμενο σημείο, όταν έχουμε αναπτυξιακά προγράμματα και την εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο, να δούμε τι θα γίνεται σε αυτή την εταιρική σχέση με βάση εθνικές αρχές όπως και με το άρθρο 12 θα είναι τότε μια πρόταση που μπορεί να υιοθετηθεί. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 12, ότι οι τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές θα πρέπει να εμπλέκονται. Και πάλι αυτό το βρίσκω εδώ λίγο λειτουργικό, όχι πολύ λειτουργικό, μάλλον αντιπαραγωγικό κιόλα για τον διάλογο για την πολιτική και τον πολιτικό διάλογο, άρθρο 13, μια παρατήρηση. Εδώ πιστεύει ο εισηγητής, λέει, ότι ο διάλογος για την πολιτική σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα με συνεννόηση σε σχέση με κάθε κράτος μέλος να διαμορφώνεται. Και εδώ τίθεται το θέμα για τη λειτουργικότητα και βιωσιμότητα. Το Κοινοβούλιο να έχει με κάθε κράτος μέλος μία επαφή και συμφωνία. Εδώ πιστεύω πάλι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από πλευράς της είναι πολύ θετική και καλύτερη. Διότι εκεί γίνεται αυτός ο διάλεκτος, διάλογος, πολιτικός διάλογος και διαμορφώνονται τα συμφέροντα των κρατών μελών και λαμβάνονται υπόψη εκεί. Στο άρθρο 14, περί τίνος πρόκειται εδώ, για την χρηματοδότηση πρόκειται. Εδώ πιστεύω και η παρατήρηση προηγούμενα έγινε ήδη, πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια κλίδα διάρθρωσης δομής του προϋπολογισμού πώς, ε, ε, εφόσον κάποια προγράμματα βρίσκονται υπό εξέλιξη. Η πρόταση στα εθνικά, για τα εθνικά αυτά προγράμματα αναφέρεται στο 2014 έως το 2020. Από το 2014 στο 2020. Συγγνώμη, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Πρέπει να βιαστούμε λίγο. Πιέζει ο χρόνος. Δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Λυπούμε που το λέω. Συγγνώμη ζητώ γι' αυτό. Πρόεδρε, λέει ο μιλητής, ολοκληρώνω στην αρχή είχαμε μια ώρα καθυστέρηση λόγω ψηφοφοριών. Τώρα αυτοί που παίρνουν τον λόγο τελευταίοι πρέπει λέει να βιάζονται και σε ελάχιστο χρόνο να ολοκληρώνουν. Πώς γίνονται όλα αυτά για το σχέδιο προϋπολογισμού, για την πρόταση προϋπολογισμού. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να έχουμε μια τέτοια διαθρωμένη πρόταση για τα κράτη-μέλη μέχρι το 2020. Εδώ υπάρχουν αιτήσιοι προϋπολογισμοί μόνο και πάλι ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο, ένα προγραμματισμένο σχέδιο πρέπει να λάβουμε υπόψη. Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες παρατηρήσεις που έχω υπόψη μου να κάνω, αλλά δεν θα τις κάνω, μια και πιέζει ο χρόνος και δεν είναι επαρκής, δεν αρκεί ο χρόνος για τον προγραμματισμό πρέπει να λειτουργεί καλά στις εργασίες της Επιτροπής μας. Πρόεδρε, παρακαλώ να ασκήσετε επιρροή στο, στη γραμματεία ώστε να εκπονεί προγράμματα συνεδριάσεων που θα είναι λειτουργικά και αποτελεσματικά. Όχι να καθυστερούμε μια ολόκληρη ώρα με κάποια άλλα θέματα και στο τέλος όταν έχουμε θέματα παρεμβάσεων προς συζήτηση να βιαζόμαστε και να τερματίζουμε προτού ολοκληρώσει κανείς. Δεν μπορεί κανείς να δουλεύει αποτελεσματικά έτσι. Σας ευχαριστούμε κύριε λέει ο Πρόεδρος. Επιμένω και εμένα όλος, όμως πρέπει να πω. Έχουμε αυτό το πρόβλημα. Τι να κάνουμε. Μια μισή ώρα ψηφίζαμε ή δύο ώρες έστω και τώρα ακόμα έχουμε τέσσερα ακόμα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Λοιπόν, θα κάθε λεπτό που έχουμε στη διάθεσή μας ε, θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε με διαρμηνία. γιατί διαφορετικά θα το μετανιώσουμε. Να βοηθήσετε γιατί έχουμε τέσσερα ακόμα σημεία και κάθε ένα από αυτά τα σημεία θεωρούν οι εισηγητές και οι σκιώδεις εισηγητές ότι είναι το πιο σημαντικό, το σημαντικότερο όλων. Να τα λάβετε αυτά όλα υπόψη, ώστε να μπορέσει να υπαρκέσει ο χρόνος. Η κυρία Κέλλερ παρακαλώ. Mm, Βλέπω να υπάρχει ακόμα ένα πρόβλημα με αυτό. Κάνει ε, κάποιες γενικές προσανατολιστικές γραμμές, γραμμές και μετά έχουμε αυτή την ε, κατάσταση. Τώρα, η αξία των προγραμμάτων Έχω κάποια προβλήματα σε σχέση με αυτό. Έχουμε ακόμα περισσότερα κονδύλια που βλέπουμε ότι πολλές φορές δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Η αξία δηλαδή δεν είναι δεδομένη με αυτόν τον τρόπο. Για την ίδια την έκθεση τώρα. Παρατηρήσεις. Συμφωνώ σε σχέση με την αξιολόγηση και το monitoring, την παρακολούθηση. Το πρόβλημα που έχω όμως είναι με την τροπολογία 30 όπου προβλέπονται κάποιες εξαιρέσεις για τον κανόνα ότι θα πρέπει να δημοσιοποιούνται, λέει όλα αυτά. Ε, δεν συμφωνώ με αυτό. Εξαιρέσει. Γιατί δεν βλέπω να υπάρχει λόγο για κάτι τέτοιο όταν πολλά πράγματα δεν είναι δημόσιου χαρακτήρα αυτή τη στιγμή. Και τελευταία παρατήρηση. Τι εννοείτε με πολιτικέ αρχέ, civic authorities. Σα ευχαριστούμε. Τώρα η Επιτροπή πάλι έχει τον λόγο για να δώσει τις τελικές της παρατηρήσεις και περνάμε στη συνέχεια στο επόμενο σημείο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να υπενθυμίσω στα μέλη της κοινοβουλευτικής σας επιτροπής ότι σαν αποτέλεσμα των συζητήσεων που ήδη διεξήχθησαν στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου καταλήξαμε σε κάποιες πληροφορίες, σε εξειδικευμένες πτυχές. Όλα αυτά έχουν διανεμηθεί, έχουν διαβιβαστεί στη γραμματεία της κοινοβουλευτικής σας επιτροπής και πιστεύω ότι πρέπει να τα έχετε στη διάθεσή σας. το θέμα για τις διάφορες ελεγκτικές αρχές αναφέρομαι στο δελτίο FISH υπαριθμό 4 για το σύστημα ελέγχου έχω Επεξηγεί τις σκέψεις και το, τις, ε, τη λογική που βρίσκεται πίσω από αυτές τις ρυθμίσεις και ιδιαίτερα σε σχέση με το άρθρο 56 για την παρατήρηση για την εταιρική σχέση και τις ε, την άμεση παρατήρηση ότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές δομές και διαρθρώσεις για κάθε τοπική περιφερειακή αρχή κτλ. Το κατανοεί πλήρως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό και γι' αυτό καθιστούμε σαφές στην πρότασή μας ότι η εταιρική σχέση θα διοργανώνεται σύμφωνα με εθνικούς κανονισμούς και πρακτικές. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο για να έχουμε επαφή με τις κρατικές αρχές κάτω από το εθνικό επίπεδο, περιφερειακό, ε, ε, δημοτικό, ιδιαίτερα όσο όσον αφορά τις ε, περιοχές και περιφέρειες που πρέπει να βρίσκονται υπό διαδικασία ένταξης και ολοκλήρωσης ε, και αυτό σε σχέση και με την τροπολογία 16 για τους κινδύνους που ε, η, συνεπάγεται η υπερβολική ακαμψία, η δισκαμψία όσον αφορά ε, την, τον προγραμματισμό. Πρέπει να υπάρχουν λεπτομέρειες και στοιχεία στα εθνικά προγράμματα και να αποφεύγουμε να είναι τόσο δίσκαμπτα αυτά και να πρέπει διαρκώς να τροποποιούνται. Λοιπόν, Φοντάνα, παρακαλώ να είσαστε πολύ σύντομος, παρακαλώ, για να εξοικονομήσουμε χρόνο. ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τις επικρίσεις ακόμα, ευχαριστώ. Καθώς και για τις ιδέες που ακούστηκαν. Εμείς ε, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε οι αρχές, οι περιφερειακές και οι τοπικές να συμμετέχουν για να δημιουργήσουν ακαμψίες. Όχι, θέλουμε να βοηθήσουν ε, το κράτος για να κάνει κάποιους ελέγχους. Γι' αυτό θέλουμε να τις εμπλέξουμε αυτές τις αρχές. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε περισσότερη γραφειοκρατία, θέλουμε πιο απλές διαδικασίες και ελπίζουμε ότι οι τοπικές αρχές μπορούν να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί αλλιώς θα είχε νόημα αυτή η πρόταση. Σε ό,τι αφορά τώρα τα άλλα σημεία και για τον προϋπολογισμό, θα κάνουμε την αξιολόγησή μας ε, για την 1η Ιουλίου 2016 ε, και θα συζητήσουμε ξανά με την Κομισιόν το σημείο αυτό για όλα τα άλλα θέματα Είμαι στη διάθεσή σας. Σίγουρα υπήρξαν κάποια προβλήματα επικοινωνίας με ορισμένους και όδες εισηγητές. Θα προσπαθήσουμε να τα επιλύσουμε το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Φοντάνα. Και τώρα, μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου, 12 η ώρα, ε, μπορείτε να υποσ... υποβάλλετε τροπολογίες. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες 10 και 11 Οκτωβρίου στην Επιτροπή. Θα θα ψηφιστεί το κείμενο το Νοέμβριο. Συμφωνούμε, προχωρούμε πολύ πολύ γρήγορα στο επόμενο σημείο. Ταμείο για το άσυλο και την ε, μετανάστευση. Η κυρία Σιλβίκη Γιώμ είναι η συγκήτρια. Να σας ε, υπενθυμίσω ότι είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Έχουμε ακόμα τέσσερα σημεία και μόνο μία ώρα στη διάθεσή μας. Σας παρακαλώ μην το ξεχνάτε γιατί ε, θα είμαι δρακόντιος Κυρία με έχετε το λόγο. Ναι, θα το έχω μονίμως υπόψη μου, Πρόεδρε. Ωραία. Λοιπόν, τηλεγραφικά απλώς θα σας πω ότι με πολύ θετική άποψη δέχτηκα την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρόλο που είναι πολύ δύσκολο να ασχοληθούμε με το Ταμείο χωρίς να μιλήσουμε για τις οριζόντιες επιπτώσεις οποίες μόλις στήξαμε. Επίσης όσον αφορά την πρόταση το ταμείο αυτό θα βελτιώσει ορισμένα θέματα στην στρατηγική ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ιδίως τους μηχανισμούς και ε, τις επίγουσες καταστάσεις και στρέφεται περισσότερο προς την επίτευξη αποτελεσμάτων. Παρουσίασα λοιπόν ε, τις τροπολογίες μου μέσα στο πνεύμα αυτό και προσπαθούμε να έχουμε ένα πιο αποτελεσματικό μέσον αλλά εάν προσπαθήσει κανείς να προσαρμοστεί μπορεί να δημιουργηθούν ανησυχίες. Γι' αυτό και αναφέρθηκα εις τις ε, πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν καλύτερες προσαρμογές. Ορισμένα θέματα επ' αυτών των τροπολογιών. Καταρχήν θέλουμε να στραφούμε προς τα αποτελέσματα και για να γίνει μία ε, αξιολόγηση των στόχων ε, προτείνω να εντείνουμε τους δείκτες οι οποίοι, τους οποίους διαθέτουμε και ιδίω τους δείκτες που επιτυγχάνουν ποιοτικό αποτέλεσμα. Το συζήτησα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι θα προχωρήσουμε. Όσον αφορά το δεύτερο στόχο των ε, τροπολογιών είναι να βελτιώσουμε τα χαρακτηριστικά του ασύλου και ιδίω του ορισμούς, διότι οι ορισμοί δεν είναι ταυτόσιμοι στα διάφορα ε, κείμενα τα οποία μας απασχολούν. Επίσης το τρίτο θα ήταν να μπορεί να μπορεί να είναι πιο... Θα ήταν δυνατόν να κλείσει το μικρόφωνο του Προέδρου γιατί υπάρχει μικροφωνισμός και είναι πρόβλημα αυτό για τους γερμηνείς. <laughs> Τέταρτο σημείο να υπάρχει μία δίκαιη κατανομή των χρηματοδοτήσεων διότι θα επανέλθω σε αυτά που είπε και ο κύριος Φοντάνα για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των κρατών μελών μόλις το ανέφερα αλλά επίσης πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά θα συνάδουν με μία δίκαιη κατανομή των πόρων. Γι' αυτό και θα ήθελα να υπάρχει ένας πιο γενικός διάλογος και ε, καλό να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και των εμπλεκομένων δημοσίων αρχών και της κοινωνίας των πολιτών και των διεθνών οργανώσεων. Είναι μια συζήτηση την οποία μόλις κάναμε. Ε, τέλος, ε, όσον αφορά την εξωτερική διάσταση των πολιτικών επ' αυτού έχω μία ανησυχία την οποία ίσως δύσκολα θα εκφράσω εδώ αλλά σας το λέω διότι τα μέτρα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν μέσω του ταμείου αυτού αναφέρονται στους εξωτερικούς στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης και στρέφονται προς τρίτες χώρες οι οποίες εμπλέκονται αλλά θα πρέπει να έχουμε επιπρόσθετα μέτρα κατά τρόπον ο διαχωρισμός αυτός των αρμοδιοτήτων και των εφαρμογών να είναι σαφής και να μην υπάρχει σύγχυση μεταξύ των χρηματοδοτήσεων. Γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρξει μια ειδική υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να επιτύχει καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών και φορέων που εμπλέκονται και όλα αυτά βέβαια αναφέρονται σε αυτό το σχέδιο κανονισμού. Και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, προτείνουμε να έχουμε πιο σαφείς κανόνες σχετικά με την την μετεγκατάσταση, ιδίω όσον αφορά τα βασικά δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα των εμπλεκομένων ατόμων και να υπάρχει μία εφαρμογή του ασύλου και της μετανάστευσης αλλά αυτό θα αναφέρεται σε μία συζήτηση πιο γενική δηλαδή να γίνει μία μεταρρύθμιση στο μέσο της διαδρομής όπως το ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τέλος το τελευταίο σημείο είναι η αλληλεγγύη. Είναι απαραίτητο για μένα το άρθρο 80 να αποτελέσει μέρος αυτής της ε, νομικής βάσεως παρόλο που αντιλαμβάνουμε μέχρι τώρα ότι είναι προβληματικό και αντί να τροποποιήσω την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είπα να δώσουμε μία διαφορετική διατύπωση βάσει του άρθρου 80 για να δώσουμε το μήνυμα στο Συμβούλιο ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε ενωμένοι στις προσπάθειές μας επιλύσεων των προβλημάτων. Ευχαριστώ. Και τώρα παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναφερθεί μόνο στα απαραίτητα σημεία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο η κυρία Πάικ. Ευχαριστώ και Κυπριακή Προεδρία. Πολύ σύντομα. Ε, σχολίασαμε το πρωί κάποια σημεία που αφορούν και αυτή την έκθεση. Καταρχάς, ε, ε, το πότε θα γίνει η διάμεση έκθεση, το θέμα των ποσοστών και όχι των ποσών. Ε, στο μέσο και επίσης την προσέγγιση που έχουμε για τους δείκτες. Δεν θα επαναλάβω αυτές τις παρατηρήσεις. Ε, καλό την εισηγείτε να σκεφτεί την ιδέα των ποιοτικών δικτών. Ξανά, καταλαβαίνουμε την αντίρρησή της, αλλά θα πρέπει να έχουμε ε, δείκτες μετρήσιμους. Κάποια άλλα θέματα που έθιξε τώρα. Καλωσορίζω την υποστήριξή της για την εταιρική σχέση. Είναι πολύ σημαντική στον τομέα που καλύπτει το Ταμείο Άσυλου και Μετανάστευσης και πιστεύω ότι θα σταλεί μήνυμα στα κράτη-μέλη που γενικά είναι απρόθυμα να θεωρήσουν ε, ότι αυτή η εταιρική σχέση δεν υπάρχει στον τομέα της ε, εσωτερικής ασφάλειας. Είναι οριζόντιο αυτό το θέμα και ελπίζουμε να μας υποστηρίξουν. Στο θέμα Τη εξωτερική ε, δράση ε, στι τρίτε χώρε Η εξωτερική διάσταση του Ταμείου είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτό αφορά και το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευση, αλλά και το τμήμα ε, της, ε, των θεωρήσεων. Είναι πολύ σημαντικό η Κομισιόν στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να εξασφαλίσει καλό συντονισμό, συμπληρωματικότητα. Ε, δεν είμαστε πεπισμένοι ότι η προσέγγιση που προτείνει η συγκήτρια είναι η καλύτερη. είναι πολύ βαριά η διαδικασία αυτή για να προωθηθεί. Ε, υποστηρίζουμε γενικά τις τροπολογίες της εισηγήτριας για την ε, επαντεκατάσταση των ατόμων. Έχουμε όμως κάποιες δυσκολίες να καταλάβουμε την προσέγγιση που έχει για τον ορισμό των μελών οικογένειας. Ε, για αυτό το σημείο και για άλλα σημεία μπορούμε να συνεχίσουμε την πολύ καλή συνεργασία με την εισηγήτρια. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Η Προεδρία θέλει να προσθέσει κάτι. Thank ε, η ίδια στρατηγική ισχύει και για τη διαχείριση της πρότασης κανονισμού για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης. Να ενημερώσω μόνο ότι μέχρι τώρα έχουν ολοκληρωθεί τρεις αναγνώσεις αυτή την πρόταση κανονισμού και η Προεδρία προτίθεται να προχωρήσει το κείμενο σε επίπεδο σύγκλησης των θέσεων και ακολούθως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης για τα ζητήματα που είναι κοινά με τον οριζόντιο κανονισμό είναι ανάγκη να υπάρχει καλός συντονισμό τόσο από μέρου του Συμβουλίου όσο και από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, τέλος, η αλληλεγγύη αποτελεί προτεραιότητα της Προεδρίας όπως δήλωσε και η υπουργό εσωτερικών ε, το πρωί και θα συζητηθεί σε αυτό το πλαίσιο στην ομάδα εργασίας. Ευελπιστούμε και εδώ σε μια πολύ καλή συνεργασία και συζήτηση με το Κοινοβούλιο και την κυρία Γκυγιό, όπου διαφαίνεται καλή πρόθεση συνεργασίας. Ευχαριστώ. Thank you. Now we got one shadow here, Mr. Tavares. You hardly had... Που είναι ισχυώδης εισηγητής. Έχετε πάρα πολύ καλούς λόγους για να συντομεύσετε. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω πορτογαλικά, Πρόεδρε. Πολύ εντάχει. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένο με τη συνεργασία σε σχέση με την εισηγήτρια Σιλβί Γκυγιόμ, συνεργασία που προσέφερε στους κοιόδη εισηγητέ για αυτό το χαρτοφυλάκιο, για αυτό το θέμα. Ήταν πολύ καλή η δουλειά που κάναμε από κοινού. Υποστηρίζω τον γενικό προσανατολισμό που ελήφθη σε σχέση με το έργο αυτό. Θα ήθελα να πω ε, όσον αφορά την Επιτροπή και το Συμβούλιο, ότι το Κοινοβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο, σε σχέση με την θέση της ομάδας μου για αυτό το θέμα του αμαλγάματος των ταμείων θα πρέπει να υπάρχει ελαστικότητα, να λαμβάνεται υπόψη αυτή η κατάσταση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μπορεί αυτό να επιτευχθεί και μπορεί να έχουμε καρποφόρο αποτέλεσμα από αυτό το αμάλγαμα, από αυτή τη σύνθεση, όταν θα είναι σαφές ότι θα έχει τον δημοκρατικό έλεγχο για τη χρήση αυτών των κονδυλίων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έχει ρόλο να διαδραματίσει σε σχέση με τι προτεραιότητε για αυτά τα κονδύλια, για αυτούς για αυτά τα ταμεία και κάποια τμήματα αυτών των ταμείων, για παράδειγμα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι είναι ερμητικά κλειστά, στεγανά κλειστά σε σχέση με τους άλλους εμπλεκόμενους. Δεν θέλω να υπάρξει καμιά αμφιβολία γι' αυτό σε σχέση με το Ταμείο ή τμήμα του Ταμείου που υποστηρίζει τις δυνατότητες επανεγκατάστασης ε, να ε, χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες επιστροφής για παράδειγμα. Για την περίοδο που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας για να καταθέσουμε τροπολογίες για αυτή την έκθεση όλοι θα πρέπει να προβληματιστούμε σε βάθος να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε πολλά από αυτά τα πράγματα. Η συγγήτρια έκανε πολλή δουλειά και οι δικές μου τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν και μόνο μέσω εχεγγύων, μέσω εγγυήσεων σαφών που θα δοθούν στις κοινοβουλευτικές επιτροπές για την επίτευξη των στόχων, μπορώ να δώσω υποστήριξη από πλευρά μου για τι προτάσει αυτέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αν δεν έχουμε άλλου σκιώδει, εσεί κύριε Μπρό, για να παρέμβετε. Ενδιαφέρει αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ταβάρες να μην έχουμε ξεχωριστά χρήματα τα οποία ενώ θα είναι για εγκατάσταση να χρησιμοποιούνται για την επιστροφή. Μου είπε η γραμματεία την προηγούμενη εβδομάδα όταν ετέθη αυτό το θέμα ότι για τις επιστροφές και επανεγκαταστάσεις τα κονδύλια βρισκόντουσαν στο ίδιο ταμείο. Ε, δεν είναι δηλαδή στεγανά και ξεχωριστά για ξεχωριστή χρήση. Δεν ξέρω αν κατάλαβα σωστά και μου τα είπαν σωστά. Συμβαίνει αυτό. Σα Σας ευχαριστώ που είσαστε τόσο σύντομος. Τώρα μπορούμε αν γίνεται να περάσουμε αμέσω στα συμπεράσματα από πλευρά τη συγγήτρια κυρία Γκυλιόμ ή αν θέλει κάποιο άλλο να παρέμβει, να κάνει κάποια σύντομα σχόλια. Όχι, κανείς. Η κυρία Γκυγιόμ λοιπόν. Μία φράση. γκυλιομ λοιπον μια αφορά του ποιοτικού δείκτε, ε, ε, ε, εγώ δεν έχω πρόβλημα για τους ποσοτικούς αλλά τους ποιοτικούς τους οποίους μπορούμε επίσης να μετρήσουμε πιο επακριβώς παρά να μιλάμε γενικώ για ποσοτικούς δείκτες όταν κοιτάζουμε και αναλύουμε τη χώρα προέλευσης, προέλευσης για τα θέματα ασύλου είναι κάτι που είναι μετρήσιμο. Όσον αφορά αφορά τον ορισμό της οικογενείας είναι μια συζήτηση την οποία κάνουμε συχνά και πιστεύω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε ένα σωστό ορισμό. Ακριβώς αυτό ήταν η κυρία Γκυγιόμ. Ευχαριστώ. Ε, για το θέμα της εκθέσεως και θέλω απλούστατα να σας πω ποια είναι η ημερομηνία ε, ε, για την προθεσμία καταθέσεω των τροπολογισμών 5 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι εντάξει τότε μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα στο 22 τα, η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία σύμφωνα και θυμάστε ότι εδώ είναι ε, ε, το θέμα του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16 Φεβρουαρίου 2012 η οποία άνοιξε το δρόμο για μία έκθεση σχετικά με το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων του, στην Ουγγαρία. Ο κύριος Ταβάρες είναι εισηγητής ο οποίος θα παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το θέμα αυτό στην Ουγγαρία. Θα ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Ταβάρες και στη συνέχεια θα γίνουν ορισμένες συζητήσεις. Πάντοτε βέβαια έχετε υπόψη σας ότι έχουμε περιορισμένο χρόνο και δίνουμε το λόγο στον κύριο Ταβάρες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τι συνέβη, τι είναι καινούριο από την τελευταία φορά που είχαμε συζήτηση για αυτό το χαρτοφυλάκιο σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επίτροπη. Το καινούριο είναι τώρα έχουμε εγκρίνει μια ad hoc αντιπροσωπεία για τη Βουδαπέστη που θα διεξαχθεί την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, από τις 24 έως 26 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία φυσικά με τις ε, Ουγγρικές Αρχές για να μπορέσει αυτή η αντιπροσωπεία να προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτή την αποστολή της. Και αποφασίσαμε ακριβώς για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε μία από τις υποσχέσεις που κάναμε στις πρώτες συζητήσεις μας, να έχουμε μία προσέγγιση που θα βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα αντικειμενικά και θα είναι δίκαια και σφαιρική ε, ολιστικής προσέγγισης για όσα συμβαίνουν στην ε, Ουγγαρία και στα οποία αναφέρεται το ψήφισμά μας στις 16 Φεβρουαρίου. Προπαρασκευή μια σειρά ε, εγγράφων εργασίας για αυτά τα γεγονότα και συμβάντα. Το πρώτο έγγραφο είναι αυτό για τις δικαστικές πτυχές, τις πτυχές του δικαστικού, της δικαστικής συνιστώσας για τα τεκτενόμενα στην Ουγγαρία. Ο συνάδελφος Έγγελ που συμφώνησε για την προετοιμασία αυτού του εγγράφου μαζί μου να εργαστεί και άλλα επίσης έγγραφα εργασίας που θα προετοιμαστούν με άλλους σκιώδεις εισηγητές από τις άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες ώστε να μπορούμε έτσι να έχουμε μια πλήρη σφαιρική εικόνα πολυσχηδή και πολυμερή και που θα καλύπτει το δυνατόν περισσότερο τις απόψεις και τις πτυχές ε, ε, και απόψεις ε, από την Επιτροπή μας. Και σε σχέση με αυτά που είπα για τον κύριο Έγκλ για την ευκαιρία για την παρουσίαση αυτών των πτυχών αυτού του εγγράφου, συσχετίζεται με δύο κύριους, ε, κύρια νομοθετήματα που εγκρίθηκαν, κύριους νόμους από την Βουλή της Ουγγαρίας για το δικαστικό σκέλος, για τη δημιουργία του εθνικού δικαστικού ε, σκέλους και για την ε, ηλικία συνταξιοδότησης δικαστών, για πιθανές πτυχές κάποιων περιπτώσεων που τίθενται υπό ε, δικαστική ε, εξέταση στην ε, Ουγγαρία για το συνταγματικό δικαστήριο την προσέγγιση αντικειμενικότητας και αμεροληψίας όσον αφορά το δικαστικό σύστημα στην Ουγγαρία. Φυσικά δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω σε κανένα ότι η ανεξαρτησία του δικαστικού σκέλους είναι ακρογωνιαίος λήθος κάθε δημοκρατικού καθεστώτος και δημοκρατίας. Ο διαχωρισμός των εξουσιών που ισχύει ως χαρακτηριστικό στοιχείο σε όλα τα κράτη-μέλη και ως ακρογωνιαίος λήθος σε όλα. Ακούσαμε και μάθαμε ότι κάποιες πτυχές ε, για τα νομοθετήματα για το δικαστικό σκέλος τροποποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο μετά από σύσταση της ε, Επιτροπής ε, και της Ευρώπης έχουν ολοκληρωθεί δηλαδή κάποιες αλλαγές που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί βέβαια στο έγγραφό μας να είσαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουμε να έχουμε όσες ε, διατυπώσεις ε, και αναδιατυπώσεις αυτού του εγγράφου θα χρειαστεί για να επικαιροποιηθεί το έγγραφο αυτό με όλες τις αλλαγές μόλις οι μεταφράσεις και τα στοιχεία θα μας έχουν διαβιβαστεί από τις Ουγγρικές Αρχές ώστε να είμαστε πλήρεις. Αυτά για αυτή τη στιγμή. Επαρκούμε σε αυτές τις παρατηρήσεις. Και ενδιαφέρομαι και προσβλέπω να ακούσω τις απόψεις των μελών και τις παρατηρήσεις σας και θα έλεγα ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε και με τον συνεισηγητή, τον κύριο Φρανκ Έγγελ, παρακαλώ. Thank you, Mr. Tavares. Πολύ σας ευχαριστούμε κύριε Ταβάρες. Ευχαριστούμε. Τώρα λοιπόν ας ανοίξει η δυνατότητα να παρέμουν τα μέλη. Ίσως εσείς πρώτος κύριε Έγκελ, συμφωνείτε. Πρώτος εσείς λοιπόν. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντιμετωπίζουμε με αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα μέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία μας για την Ουγγαρία στα πλαίσια της έκθεσης. Ε, κάτι που μας ανέθεσε η Ολομέλεια. Ξεκινήσαμε να προετοιμάζουμε ένα έγγραφο για το δικαστικό σύστημα. Θα ακολουθήσουν κι άλλα με τις κλασικές ε, κοινοβουλευτικές προθεσμίες, γιατί θα πρέπει να μεταφραστεί, υπάρχουν μια σειρά από πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και καθώς εμείς ετοιμάζουμε το έγγραφο και μεταφράζεται το έγγραφο, παράλληλα οι ουγγρικές αρχές, όπως συμβαίνει συχνά, ήταν σε μόνιμη επαφή με την Επιτροπή της Βενετίας σε αυτή την περίπτωση για να δουν τι έπρεπε τελικά να εφαρμόσουν ως νομοθετικές αλλαγές. Και τελικά έγινε στις 2 Ιουλίου ε, η ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο ε, πριν από μια εβδομάδα δηλαδή. Έχουμε ένα έγγραφο λοιπόν, το οποίο είναι κάτι λιγότερο από αυτό που θα έπρεπε να είναι όταν εμείς είχαμε σκεφτεί να το συντάξουμε και τελικά θα πρέπει να το αλλάξουμε. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή που είναι στη διάθεσή μας να συνεισφέρει και αυτός. Τον ευχαριστώ που επίσης είπε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες εκδοχές του κειμένου, γιατί αυτό το έγγραφο δεν είναι ολοκληρωμένο, δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Ποια. Είπαμε στην αρχή ότι αυτά τα κείμενα είχαν σαν σκοπό να αποτελέσουν ένα checklist. Δηλαδή, όταν πηγαίνουμε στην Ουγγαρία και μιλάμε με τις Ουγγρικές Αρχές, γνωρίζουμε τις επικρίσεις που έχουν αναφερθεί για τις συνταγματικές και δικαστικές διατάξεις στην Ουγγαρία, νομικές διατάξεις και ανάλογα με αυτά κάνουμε προτάσεις για να αλλάξει η Ουγγαρία τα συγκεκριμένα σημεία. Είναι μια συνεχής διαδικασία. Έτσι, το περιμέναμε κιόλας. Και οι δικές μας προθεσμίες, τα δικά μας ορόσημα, μας φέρνουν σε δύσκολη θέση. Ε, αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο και αν συνεχιστεί έτσι επί μακρόν αυτή η κατάσταση. Επί της ουσίας τώρα του εγγράφου θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις πιο πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές της Ουγγαρίας στην εικόνα που αποτυπώνουμε. Και αυτό θα είναι η βάση των συζητήσεων που θα κάνουμε στην Ουγγαρία το Σεπτέμβριο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η διαδικασία δεν θα έχει ολοκληρωθεί. Μου είπαν, α πούμε, ότι το θέμα τη ε, ηλικία ταξιδότηση των δικαστών εξετάζεται ξανά και ξανά. Δεν έχει ρυθμιστεί με την ε, τελευταία ε, νομοθεσία που πέρασε στη Βουδαπέστη. Α, είναι σε φάση ακόμα συζήτηση λοιπόν. Δεν έχει οριστικοποιηθεί και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο σε πραγματικό χρόνο να απεικονίζουμε τις εξελίξεις και τις αλλαγές. Και τώρα να, να επανέλθω σε κάτι που είπα την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Δεδομένου ότι οι Ουγγρικές Αρχές από την αρχή ήταν διατεθειμένες ε, να κάνουν αυτέ τι αλλαγέ που τους προτείναμε και κάναν μεγάλε προσπάθειε ούτω ώστε να εφαρμόσουν τι νομοθετικέ αλλαγέ που περιμένουμε από αυτέ. Και μια και είναι μια διαδικασία η οποία δεν θα είναι αέναη, είναι μια διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί τους επόμενους ε, μήνες και όχι χρόνια. Γι' αυτό πρέπει να κοιτάξουμε και το δικό μας χρονοδιάγραμμα, τις δικές μας προθεσμίες. Γιατί αν εμείς καθυστερήσουμε πολύ, μπορεί τελικά να καταλήξουμε μια έκθεση για την κατάσταση στην Ουγγαρία που δεν θα απεικονίζει την τότε κατάσταση. Δηλαδή δεν θα είμαστε επίκαιροι. Δεν, ενδιαφέρει, δεν θα ενδιαφέρει τότε η έκθεσή μας ούτε την Επιτροπή αυτή. Ούτε κανέναν. Επομένω, το πρώτο που πρέπει να πω για το έγγραφο είναι ότι θα πρέπει να το εμπλουτίσουμε για να λάβουμε υπόψη όλα τα στοιχεία και πρέπει να συμφωνήσουμε επί ενός χρονοδιαγράμματος που θα μας επιτρέπει να ολοκληρώσουμε με μια ταχύτητα που να μην είναι κατώτερη από αυτή με την οποία λειτουργούν ουγγρικές αρχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κάποιον είδα να θέλει το λόγο, τον κύριο Μπρόγκς και ποιον άλλον, την κυρία Ίντεβελτ. Πρώτα κυρία Ιντβελτ και μετά ο κύριος Μπρόνξ. Όπως θέλετε. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους εισηγητές για τη δουλειά που κάνανε και για την επιλογή της μεθόδου. Η όλη κατάσταση δείχνει ξεκάθαρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τα κατάλληλα μέσα για να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να έτσι στα ψαχτά να βρούμε την κατάλληλη μέθοδο. Και η μέθοδος που έχετε επιλέξει είναι πολύ λογική. Μένετε στα γεγονότα και δημιουργείτε, και δημιουργείτε με αυτόν τον τρόπο που δουλεύετε την απαραίτητη νυφαλιότητα που χρειάζεται για να κοιτάξουμε αυτά τα θέματα, ίσως και άλλα θέματα. Όταν υιοθετήσουμε την έκθεση θα μπορούσαμε λοιπόν να αξιολογήσουμε το πώς λειτουργεί ως μέσο για έλεγχο της κατάστασης στα κράτη-μέλη. Γιατί θεωρώ ότι και άλλα κράτη-μέλη, και το δικό μου δεν αποκλείεται, ίσως και το δικό μου κράτος μέλος, θα πρέπει να το ελέγξουμε εκ του σύνεγγυς. Μία ερώτηση έχω ουσιαστικά και δεν ξέρω αν μπορείτε να την απαντήσετε. Άκουσα μια ιστορία, αλλά δεν έχω ιδέα αν είναι αληθινή, ότι την περασμένη εβδομάδα ή πριν από δύο εβδομάδες ένας δικαστής απολύθηκε. Ένας γνωστός δικαστής που ήταν πολύ επικριτικός απέναντι στην κυβέρνηση. Δεν έχει καμία σχέση αυτό δηλαδή με τους νόμους που έχουν περάσει, αλλά περισσότερο με την πρακτική, με τον τρόπο που εφαρμόζονται και με τους πιθανούς κινδύνους. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό που έμαθα, αυτό που σας λέω. I mean, I mean, <laughs> Mrs. Guns or Mrs κυρία Γκάνση, κυρία Γκάλ. Ποια από τις δύο θέλει να απαντήσει πρώτη σε αυτή την ερώτηση. Και οι δύο Ουγγαρέζες ε, συνάδελφοι θα μπορούσαν να απαντήσουν πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Μπρόγκς. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Θα ήθελα να συζητήσουμε περισσότερο άλλα θέματα. Είναι αλήθεια αυτό που ακούσατε, κυρία Ιντβέλτ θα ήθελα να μιλήσω περισσότερο αυτά που είπε ο κ. Σέγγελ, ότι είναι μια ενεξελίξη διαδικασία στην Ουγγαρία. Όταν ήταν στο Λομέλιο ο Πρωθυπουργό, ε, περήφανα ανέφερε ότι διάφοροι νόμοι α, υιοθετήθηκαν στην Ουγγαρία μέσα σε ένα χρόνο. Ε, όχι μόνο εμεί δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ταχύτητά τους, αλλά και οι Ούγγροι ε, δικηγόροι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα τεκτενόμενα ε, σε νομοθετικό επίπεδο στην Ουγγαρία. Αυτό που συζητήσαμε νωρίτερα είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό να πάμε στην Ουγγαρία, να επισκεφτούμε τη χώρα, να δούμε όλες αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Γιατί ένα είναι το νομοθετικό στοιχείο του προβλήματος, αλλά άλλο πολύ σημαντικό είναι να δούμε τις επιπτώσεις. Να δούμε την διαδικασία εφαρμογής επιτόπου. Δεν νομίζω ότι έχουμε χρόνο να μπούμε σε λεπτομέρειες. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό να πάμε στην Ουγγαρία για να δούμε τι γίνεται πραγματικά. Ευχαριστώ. Για να ολοκληρώσουμε αυτή την απάντηση, η κυρία Γκάλ και μετά ο κύριος Μπρόγκς. Δεν ξέρω τι συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτό που ξέρω είναι ότι και λόγω της αλλαγής που πέρασε στις 2 Ιουλίου, όταν λαμβάνεται μια απόφαση υπάρχει δυνατότητα να πάει κανείς με την απόφαση στο δικαστήριο. Αυτό αναφέρεται σαφώς. Με τις νέες αλλαγές που πέρασαν, με τις νέες τροπολογίες. Ούτως ή άλλως το θέμα αυτό το εξετάζει το συνταγματικό δικαστήριο και αυτό δείχνει ότι ναι, τα... οι θεσμοί λειτουργούν στην Ουγγαρία. Συμφωνώ επίσης με τον κύριο Έγγελ ότι είναι σημαντικό να δούμε τι άλλαξε και τι οθετήθηκε στα πλαίσια όλης αυτής της διαδικασίας. Αν κοιτάξετε τι συνέβη σε άλλα κρατημέλη, τελικά ελπίζω να μην στυλιτεύσετε την Ουγγαρία ως χειρότερη υπόθεση, ως τη χειρότερη χώρα, όπως συνέβη τους τελευταίους μήνες είναι επιθυμητό για τη μέθοδο διορισμού και τη μονιμότητα των δικαστών να ενθαρρύνουμε την ανεξαρτησία τους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο πάντως, μέχρι το 2006, ε, όταν δημιουργήθηκε η Δικαστική Επιτροπή, ο διορισμός των δικαστών ε, ήταν θέμα των πολιτικών και του ε, Υπουργού Δικαιοσύνης, παρότι υπήρχαν κάποιες άτυπες διαβουλεύσεις. Ε, και πολλοί από τους σημερινούς δικαστές διορίστηκαν με το παλιό ε, δικαστικό σύστημα που εξηγεί εν μέρη ε, κάποιες περίεργες αποφάσεις σε ορισμένες δικαστικές υποθέσεις. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το πώς θα συμπεριφέρονται οι, δικαστές σε πολλές χώρες που δεν εκφράζονται ελεύθερα και δεν διορίζονται με τις πιο αυστηρές διαδικασίες. Επίσης δεν δείχνουν δεν θέλω να υπερασπιστώ την ε, Ουγγαρία, αλλά πριν τη στυλιτέσουμε θα πρέπει ο καθένα θα πρέπει να εξετάσει το πώ λειτουργούν οι δικαστέ στη δική του χώρα. Ε, κύριε Ταβάρη, ε, σε εσά δίνω το λόγο για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση προ το παρόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και γι' αυτό το τμήμα των υποεξέλιξης συζητήσεων για την Ουγγαρία, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σημειώνω όλα τα σχόλια που ακούστηκαν. Ήθελα μόνο να πω ότι το ότι δεν είναι επικαιροποιημένο αυτό το έγγραφο δεν είναι κάτι αμετάκλητο ως κατάσταση. Φυσικά με τις τελευταίες πληροφορίες που είχαμε από την Ουγγαρία είχε συνταθεί και αυτά τα πράγματα αλλάζουν βέβαια. Και βρίσκεται υπό εξέλιξη η κατάσταση. Για αυτή την παρατήρηση αυτό ακριβώς κάνουμε και αντιμετωπίζουμε. Κάθε έκθεση σε αυτό το σώμα βρίσκεται υπό αυτό το πρίσμα αξιολογούμε, παρακολουθούμε μια κατάσταση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, το κράτος δικαίου της ένομης τάξης σε μια χώρα όπως την Ουγγαρία. Είναι φυσικό και φυσιολογικό να αλλάζουν κάποια πράγματα, να έχουμε θετικές ειδήσει, καλά μαντάτα ή όχι τόσο καλά μαντάτα. Και είναι πολύ δύσκολο να τηρεί κανείς το ρυθμό αυτό και να καλύπτει όλες τις πληροφορίες όπως έρχονται από αυτή τη χώρα, από την Ουγγαρία, νομοθετήματα, διαδικασίες, διεργασίες από το Κοινοβούλιο και από τα σώματα, όπως σε σχέση με την ασφάλεια, για παράδειγμα, που πρόσφατα ε, ε υπέπεσαν στην προσοχή μου. Ζητώ τα μέλη, οποιαδήποτε πληροφορία έχουν να μου τη διαβιβάσουν. Είναι ανοιχτή φυσικά η θύρα μου, η πόρτα μου για συζητήσεις για αυτό το χαρτοφυλάκιο μαζί σας. Όσο αφορά το χρονοδιάγραμμα, θα έλεγα έχουμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο άμεσο μέλλον, που είναι η αποστολή μας. Αυτό το έγγραφο εργασίας και τα άλλα που θα προετοιμαστούν στο άμεσο μέλλον είναι προκαταρκτικές, προπαρασκευαστικές σημειώσεις για μετά από τις θερινές διακοπές. Όταν θα έρθουμε, θα επιστρέψουμε από την Ουγγαρία, θα έχουμε συναγάγει κάποια συμπεράσματα, θα έχουμε καταλήξει σε ένα πιο καθοριστικό πλαίσιο, όσο το δυνατόν γίνεται πιο καθοριστικό στη διατυπώσεις και όλα αυτά τα στοιχεία έγγραφα με τους σκιώδεις εισηγητές και τις κοινοβουλευτικές ομάδες από κοινού θα διασφαλίσουν οι παρεμβάσεις και οι συνεισφορές και εκείνων των κοινοβουλευτικών ομάδων που επιθυμούν να ληφθούν υπόψη θα αποτελέσουν τη βάση της ε, εργασίας ε, για τη σύνταξη αυτών των ε, εκθέσεων, αυτών των στοιχείων. Αυτό είναι το modus operandi, ο τρόπος εργασίας και προσέγγισης από πλευράς μας. Τουλάχιστον για το προβλέψιμο μέλλον, μια και πρόκειται για μια συνενετική και από κοινού προσπάθεια και διεργασία. Θα ήθελα να πω για να ολοκληρώσω, μόνο δύο παρατηρήσεις θα είχα για την Επιτροπή Βενετία στην Venice Commission όπως ε, αναφέρθηκε εδώ, οι τελευταίες αλλαγές όσον αφορά την νομοθεσία σε σχέση με το δικαστικό στην Ουγγαρία έγιναν ανταποκρινόμενοι στα σχόλια και τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Βενετίας. Υπήρξε μια πολύ καλή έκθεση που συντάχθηκε από την Επιτροπή Βενετίας ε, που όλοι θεωρούμε εδώ ως πρότυπο, υπόδειγμα για την αξιολόγηση των δικαστικών ε, θεμάτων και του δικαστικού σκέλους στην Ουγγαρία. Έχουμε αντλήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στοιχεία από την έκθεση της Επιτροπής Βενετίας και μια και αυτό που κάνουμε και έχουμε ε, μέγιστο ενδιαφέρον για τις απόψεις και τις ε, τοποθετήσεις αυτής της Επιτροπής Βενετίας για τα νομοθετήματα και τις αλλαγές σε σχέση με την Ουγγαρία. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση. δεύτερη παρατήρηση, πρωτού ολοκληρώσω. Αναφέρθηκε σε αυτή τη συζήτηση και το θέμα άλλων κρατών μελών. Αυτό που συζητάμε όμως εδώ φυσικά είναι η περίπτωση της Ουγγαρίας. Όμως έχει και τεράστια σημασία αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή και ευρύτερα το Ευρωκοινοβούλιο να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τα τεκτενόμενα σε άλλα κράτη-μέλη. Είναι εξίσου σημαντικό να το κάνουμε με την ίδια ενεργητικότητα και αφοσίωση όπως στην περίπτωση της Ουγγαρίας και, όπως, και ως εισηγητής σε σχέση με την περίπτωση της Ουγγαρίας αλλά και ως μέλος αυτής της Επιτροπής θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μην επιτρέψουμε εμείς να παρεκκλίνουμε και να θεωρηθούμε ύποπτοι για οποιαδήποτε μεροληψία ή ιδιοτέλεια ή παρέκκληση από τις αρχές αμεροληψίας και αντικειμενικότητας. Είναι κοινέ αρχέ και αξίε που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα δικαιώματα του ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασιστείτε πάνω μου και πιστέψτε με και ομιλώ και εξ ονόματο των σκιωδών εισηγητών για αυτό το χαρτοφυλάκιο. Όλοι μα θα παρακολουθήσουμε και τι άλλε περιπτώσει όπω και τη Ουγγαρία με την ίδια ενεργητικότητα και αφοσίωση και προσοχή. Σα ευχαριστώ όλου σα. Και όπω είπα, είμαι πάντα στη διάθεσή σα πρόθυμο να συνεισφέρω σε οποιαδήποτε παρέμβαση πρόταση μελών αυτής της κοινοβουλευτική Επιτροπής του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο μέχρι ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες μας απόψε και έχουμε δύο ακόμα σημεία που αφορούν τον συνάδελφό μας κύριο Σαλβατόρη Γιακολίνο ως εισηγητή. Το πρώτο αφορά τον Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οικονομικό έτος 2013, όλα τα τμήματα. Είμαστε εδώ λοιπόν παρόντες να ακούσουμε την παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης και για τις τροπολογίες για τον προϋπολογισμό 2013 του οικονομικού έτους από τον κύριο Γιακολίνο. Θα ακούσουμε τα σχετικά από τον ίδιο, τον κύριο Γιακολίνο, και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυπριακή Προεδρία όταν, αν έχουν κάποια σύντομα σχόλια. Να θυμόσαστε, πρέπει να είναι σύντομα τα σχόλιά σας, ώστε να θέσουμε προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. Ο κύριος Ευρωβουλευτής Γιακολίνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι συντομότατος, λακωνικότατος, δεδομένου ότι είναι πολύ αργά. Ξεκινάμε με αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης για τον προϋπολογισμό του 2013, που είναι μια σημαντική χρονιά. Ε, δεδομένου ότι από το 2014 αρχίζουν οι νέε δημοσιονομικέ προοπτικέ. Επομένω, πρέπει να δούμε τι περιέχει αυτό ο προπολογισμό. Με δεδομένο το χρονικό ορίζοντα τον πολιετή 2014-2020. Τι προσπαθήσαμε να κάνουμε. Προσπαθήσαμε, και το είπαμε και στην Ολομέλη την περασμένη εβδομάδα, όταν έγινε η συζήτηση ε, για, τον για την εντολή για τον τριμερή για τον ε, διάλογο για τον προπολογισμό του 2013 ότι δεν ήμασταν ε, σύμφωνοι με κάποιες περικοπές που πρότεινε η Κομισιόν. Θα ξεκινήσω με μία περικοπή που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και που αφορά το, τα προγράμματα κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μην ξεχνάτε εξάρτητα, ότι αποφάσισε να δημιουργήσει μία επιτροπή με ειδικό καθήκον να δώσει πολιτικές κατευθύνσεις ε, και ένα κατάλογο προτεραιοτήτων, τόσο ώστε να καταπολεμήσουμε πιο αποτελεσματικά το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και, την, και το ξέπλυμα χρήματος. Ε, πρότεινα λοιπόν μια διόρθωση, μια αύξηση προφανώς. Όπως πρότεινα αύξηση σε ορισμένες άλλες παρεμβάσεις που αφορούν τα εξωτερικά σύνορα, το Ταμείο για την, ε, τον Επαναπατρισμό, το ΣΥΣ 2 με ένα αποθεματικό του 20% των πιστώσεων για την Europol, για την EASO και για την Eurojust. Πρόκειται για ένα σχέδιο που διαρθρώνεται σε διάφορα σημεία που έχει σαν στόχο να μειώσει κάποιες μειώσεις, να μειώσει κάποιες μειώσεις που επέφερε η Κομισιόν, έτσι, σε κάποιους ευαίσθητους τομείς και σε κάποιες σημαντικές δραστηριότητες που είναι τμήμα του χώρου ε, ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας, ξεκινώντας με το ρόλο των διαφόρων οργανισμών. Επίσης, κυκλοφορήσαμε ένα σχέδιο μαζί με τη Γραμματεία που αναφέρει τα όσα προτείνουμε, που σε μεγάλο βαθμό σας ανέφερε εδώ στην παρέμβασή μου. Και ανέφερα βεβαίως και στην Ολομέλεια για τη συζήτηση που έγινε για τον προϋπολογισμό του 2013 την περασμένη εβδομάδα. Επίσης, στις 26 Ιουνίου ε, ετοιμάσαμε και αυτή την έκθεση, την οποία συμπληρώσαμε και σημειώσαμε με αυτές τις ειδικέ δικές μου α, παρεμβάσεις. Το Συμβούλιο προέβλεψε περικοπές του προπολογισμού 50 εκατομμύρια και άλλες παρεμβάσεις για το ΣΥΣ2. Για το Σέγγεν θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δεδομένων των θέσεων του Συμβουλίου ότι θα πρέπει να βάλουμε σε αποθεματικό το προϋπολογισμό που προβλέπεται για το μηχανισμό αξιολόγησης του Σέγγεν. Αυτό είναι ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα που στέλνουμε, που θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για να βελτιώσουμε τις σχέσεις με το Συμβούλιο. Και ενδεχομένως να γίνει μια αναθεώρηση αυτής της απόφασης που δημιούργησε την νομοθετική βάση πρόσφατα και που τη μετέτρεψε, που τη μετέφερε μάλλον από, την, από το άρθρο 76 στο άρθρο 70, όπου το κοινοβούλιο αντιτάχθηκε. Δηλαδή δεν θέλουμε να περάσουμε από το 76 που ήταν στην απόφαση στο 70. Αυτά, Πρόεδρε, θα σταματήσω εδώ για να ακούσω τώρα τις επόμενες παρεμβάσεις. Ευχαριστώ κύριε Γιακολίνο. Η Κομισιόν σύντομα, σύντομο σχόλιο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Θέλει να πάρει το λόγο. Θέλετε να σχολιάσετε. Όχι, δεν χρειάζεται. Πολύ ωραία. Άλλα σχόλια από τους Ευρωβουλευτές. Η κυρία Κέλλερ. Έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ. Έχω μια γενική παρατήρηση, διότι μιλήσατε για το Σέγγεν και νομίζω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες αποφάσισαν να μπλοκάρουν ορισμένα θέματα στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και αυτό είναι θέμα του προπολογισμού 2013 και δεν βλέπω αυτό να αντικατοπτρίζεται ακόμη στις τροπολογίες. Πιστεύω όμως ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε ορισμένες τροπολογίες που θα δείξουν σαφώς ότι δεν δεχόμαστε τις θέσεις του Συμβουλίου και θα μπλοκάρουμε τα πράγματα εάν δεν υπάρχουν σημαντικά ποσά στο αποθεματικό. Και αυτό Αυτά θα είναι ε, τα σημεία τα οποία θα προωθήσουμε τις τελευταίες ημέρες πριν από το τέλος της προθεσμίας υποβολής των τροπολογιών. Ε, σας ευχαριστώ λέει η κυρία Γκέντς. Ε, σαν συνεισηγήτρια ήθελα να σας πω ότι η συζήτηση συνεχίζεται σχετικά με το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού για το 2013 σχετικά με τις εσωτερικές υποθέσεις και υπάρχουν ακόμη ερωτηματικά ε, ε, ε, σχετικά με τη σημασία του τομέα αυτού δηλαδή ε, εάν θα υπάρχουν περισσότερες δεσμεύσεις που να τονίζουν τις ευθύνες μας στον τομείο αυτό. Δεν ξέρουμε ε, εάν το Συμβούλιο προτίθεται να αυξήσει τον προπολογισμό και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε ένα χειρό μήνυμα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα διότι η Ευρώπη ε, πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Χρειαζόμαστε πόρους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα θέματα που εκκρεμούν και μεγαλύτερη δικαστική συνεργασία, σύγκληση των νομικών συστημάτων, εκπαίδευση της αστυνομίας και απάντηση στις διάφορες προκλήσεις. Χρειαζόμαστε δηλαδή να έχουμε αρκετή χρηματοδότηση και ένα άλλο θέμα το οποίο είχα αναφέρει προηγουμένως είναι ότι πάντοτε υπάρχει μία ανισορροπία μεταξύ των διαφόρων ταμείων εσωτερικών υποθέσεων σε σχέση με τα εξωτερικά σύνορα και δεν δίδονται επαρκή πόρη, επαρκή σπόρη στο, για τη χρηματοδότηση του θέματος των προσφύγων. Οπότε πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις για να προωθηθούν τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Αν δεν έχετε άλλα σχόλια, τότε δίνω το λόγο πάλι στον κύριο Γιακολίνο. Για το θέμα του Σέγγεντ. υπάρχει δυνατότητα ενός αποθεματικού. Καλό θα ήταν να δοθεί αυτό το σημαντικό πολιτικό μήνυμα. Όλοι είμαστε πεπισμένοι ότι το Συμβούλιο έχει διαπράξει ένα σοβαρότατο λάθος να θεωρήσει την νομοθετική βάση είναι μια διαφορετική και όχι αυτή που αφορά τη συναπόφαση για το μηχανισμό αξιολόγηση του Σέγγεν και επομένως αυτό το θέμα θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και θα δούμε τους τρόπους με τους οποίους θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε αυτό το θεματικό. Για τα άλλα θέματα, για τα θεμελιώδη δικαιώματα, για τη συνεργασία, τη δικαστική, για το θέμα της επανεγκατάστασης των μεταναστών, Αυτά τα συγκεκριμένα θέματα τα λαμβάνουμε δεόντως υπόψη στην γνωμοδότηση με τη διατύπωση που έχουμε επιλέξει, η οποία εγκρίθηκε και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Βεβαίως, ξέρετε πολύ καλά ότι χαρακτηρίζεται ο προπολογισμό από το κλίμα αυτό λιτότητας και δημοσιονομικής εξυγίανσης. Η Κομισιόν δεν σχολίασε την πιθανή τροπολογία, τις τροπολογίες δηλαδή που προτείνουμε εμείς. Ελπίζουμε, ήλπιζα τουλάχιστον, να συμμεριστεί τις προτάσεις μας. Ευχαριστούμε κύριε Γιακολίνο. Για τις τροπολογίες, μια ανακοίνωση. Μην ξεχνάτε το χρονικό περιθώριο. Η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες μπορεί να εθμιστεί στις 27 Αυγούστου 12 η ώρα. Αν δεν υπάρχετε αντιρρήσεις, να υποβληθούν στα αγγλικά παρακαλώ, ούτω ώστε να γλιτώσουμε τις μεταφράσεις. Λόγω σφιχτού χρονοδιαγράμματος, για να μπορέσουμε να είμαστε εμπρόθεσμοι. Αν δεν έχετε αντίρρηση λοιπόν, να υποβάλλετε τις τροπολογίες στα αγγλικά. Και η προθεσμία είναι 27η Αυγούστου μέχρι το μεσημέρι. Συμφωνείτε? Πολύ ωραία. Η ψηφοφορία θα γίνει λοιπόν το Σεπτέμβριο στις 3 Σεπτεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα. Πάμε στο τελευταίο σημείο. Σημείο επίσης του για Κολίνο, Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, Αστυνομική Συνεργασία, Πρόληψη και Καταπολέμηση του Εγκλήματος και Διαχείριση των Κρίσεων είναι σχέδιο έκθεσης ε, για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, Νομική Συνεργασία, Πρόληψη και Καταπολέμηση του Εγκλήματο, επαναλαμβάνει ο Πρόεδρος. Θα ακούσουμε τον εισηγητή, ίσως μπορούμε να ακούσουμε και λίγο την Επιτροπή και την Προεδρία, αν το επιθυμούν. Και αυτά θα είναι τα τελευταία λόγια πριν από τι καλοκαιρινέ διακοπέ. Κύριε Γιακολίνο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε είναι το τελευταίο θέμα της ε, σημερινής ημέρας. Φαντάζομαι ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο, σε μια στιγμή όπου το κατόφλι προσοχή σας είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Είναι ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό μέσο. Ήδη συζητήθηκε σε προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Εγώ παρουσίασα μια έκθεση τις περασμένες ε, τις προηγούμενες μέρες που συνοψίζει, που θέλω να συνοψίσω τώρα. Είναι η δυνατότητα για αστυνομική συνεργασία, πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος. Είναι πολύ σημαντικό σημείο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και τα, των αδικημάτων διασυνοριακού χαρακτήρα. Είναι καινοτόμο, ευέλικτο, ε, προστατεύουν την νόμιμη οικονομία και την, ε, τις νόμιμες επιχειρήσεις. Ε, καταπολεμούν την ανακύκλωση και τα, την ανακύκλωση του χρήματος και τα έσοδα από εγκληματικέ δραστηριότητε σε περίπτωση που έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Έχουμε κάποιου ορισμού. Να ξεκινήσω με τον ορισμό τη οργανωμένη εγκληματικότητα, όπου όπω προβλέπεται και σε άλλα νομοθετήματα είναι η άσκηση εκφοβισμού Ξαναμιλήσαμε για την έννοια των κρίσιμων υποδομών επίσης, κρίσιμες υποδομές. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε αντικειμενικούς δείχτες, ποσοτικούς, για να υλοποιήσουμε την υλοποίηση των συγκεκριμένων στόχων. Φερρυπίν να δούμε πόσες επιχειρήσεις διασυνοριακού χαρακτήρα έχουμε. Να μιλήσουμε καταρχάς και το ποσοστό του προσωπικού που συμμετέχει σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Ε, και επίσης ποιοι συμμετέχουν σε δραστηριότητες κατάρτισης. Θεωρούμε ότι η κατανομή των πόρων είναι, πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο για την πρόληψη και τη συνεργασία για την οποία μιλάμε, διαφωνώντας με την Κομισιόν, που θέλει να κατανείμουμε διαφορετικά τους πόρους αναδράση. Στο άρθρο 5, με την ε, τροπολογία 52, θέλουμε το 40% των πόρων να πάει σε δράσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Κομισιόν και το 60% δηλαδή μέσα να πηγαίνει σε προγράμματα εθνικού χαρακτήρα, ούτω ώστε να έχουμε μια μεγαλύτερη εμπλοκή των κρατών μελών, τα οποία όμως θα πρέπει να έχουν μια πιο ευέλικτη δυνατότητα χρήσης των πόρων που έχουν στη διάθεσή τους. Ταυτόχρονα θέλουμε διαφορετική κατανομή των πόρων που πηγαίνουν σε εθνικά προγράμματα με μια διανομή που θα λαμβάνει υπόψη κριτήρια τα οποία έχουμε αναδιατυπώσει σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε μια περίπτωση έχουμε διαγράψει την αναφορά στις κρίσιμες υποδομές. Έχουμε επίσης αναδιατυπώσει κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τα κράτη-μέλη που είναι υπερεκτεθειμένα σε πιέσεις μεταναστευτικές. Επίσης, τέλος, θεωρούμε ότι η αναφορά στο κεκτημένο Σέγγεν είναι ακατάλληλο, ανακατάλληλες και ανεπαρκής, γι' αυτό τις διαγράψαμε. Αυτά, εν συντομία, Πρόεδρε. Αυτά ήταν το αντικείμενο της παρέμβασης που ήθελα να κάνω για το συγκεκριμένο θέμα. Και αν έχετε περισσότερες ε, συνεισφορές, ε, είμαι στη διάθεσή σας ή οποιασδήποτε βελτιώσεις να κάνετε. Ευχαριστώ κύριε Γιακολίνο για την παρουσίαση αυτής της έκθεσης για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή το αφήσαμε τελευταίο, σημαίνει λιγότερο σημαντικό, έτσι. Last but not least, λέει και αγγλιστή ο πρόεδρος. Ας ακούσουμε τώρα κάτι σημαντικό, την Κομισιόν και την Προεδρία του Συμβουλίου. Η Κομισιόν. Θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για την έκθεσή του που ακολουθεί την ορθή κατεύθυνση και αντανακλά και μια ολόκληρη σειρά θεμάτων και ζητημάτων που εθίγησαν και από πλευρά Συμβουλίου. Και πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει και στις συζητήσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Ήδη ανέφερα αρκετές φορές στο παρελθόν τα μέσα και σε σχέση με τα μέσα αυτά θα συνεχιστεί το έργο για κοινού ε, δείκτες ε, σε workshop, ε, σε σεμινάριο για κάθε ένα από τα μέσα αυτά και το Ευρωκοινοβούλιο φυσικά και τα κράτη-μέλη προσκαλούνται να συμμετάσχουν. Με αυτή την αφορμή θα μπορέσουμε να δούμε τους κοινού δείκτες σε λεπτομέρειες. Μπορώ να επαληθεύσω και να επιβεβαιώσω ότι συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν πρόκειται για ένα ε, συναφές με το Σέγγεν ε, μέσο και γι' αυτό συμφωνούμε με την απάλληψη, διαγραφή των αναφορών σε σχέση με τις χώρες, ε, σε σχέση με αυτά τα πράγματα. Τώρα, για μια κεντρική διαχείριση όπως γνωρίζουμε είναι ένας τομέας πολιτικής αυτός που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ένα πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση εθνικών προγραμμάτων από τα κράτη-μέλη το βίωμα και η πείρα σε σχέση με εθνικό προγραμματισμό είναι πολύ πιο αποδυναμωμένη σε σχέση με άλλους τομείς ε, που αφορούν τις εσωτερικές υποθέσεις. Γι' αυτό προτείνουμε συγχρηματοδότηση 50-50 όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τη συζήτηση για τη χρηματοδότηση για τα προγράμματα προσωπικών δεδομένων ταξιδιωτών PNR έχουν υπάρξει συζητήσεις για την αύξηση του ποσοστού του ISF, αυτού του μέσου που θα αποτελεί τμήμα συνδιαχείρισης. Αυτό είναι τμήμα των συζητήσεων που βρίσκονται υπό εξέλιξη παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα θέματα, βρίσκεται υπάρχει λογική σε αυτήν την προσέγγιση. Θέτει το θέμα για τα κριτήρια κατανομής ο εισηγητή για τα κονδύλια αυτού του ταμείου. Αναφέρθηκα αρκετέ φορέ σήμερα για το δελτίο πληροφόρηση FISH σε σχέση με διάφορε πτυχέ αυτού του μέσου. Ιδιαίτερα το δελτίο FISH 2 για την κατανομή κονδυλίων χρηματοδότησης και έχουμε επεξηγήσει το πώς ακολουθούν οι ε, διαδικασίες για τα κριτήρια κατανομής. Τώρα αναφέρω αυτό γιατί υπάρχει διαφορετική κατάσταση για το Ταμείο Μετανάστευσης και Ασύλου σε σχέση με το Ταμείο για τη Διαχείριση των Συνόρων και τους ελέγχους ε, λοιπά Η προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί λοιπόν σε σχέση με αυτό το ταμείο συγκεκριμένα είναι να δούμε με τρεις αντικειμενικά κριτήρια όπως περιγράφονται που πρέπει να προστατεύονται και αυτή είναι η προσέγγιση η φιλοσοφία που μας εμπνέει. Δεν υπάρχει μονοπόλιο βέβαια σοφίας ή γνώσης και σε σχέση με τα εξωτερικά σύνορα ή θαλάσσια σύνορα για αυτό το ταμείο είναι πολύ γνωστό και κατανοούμε ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την κατανομή κονδυλίων ISF όσον αφορά τα σύνορα και θεωρήσεις διαβατηρίων. Και είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις μεταναστευτικές πιέσεις. Ωστόσο δεν είναι ο πρωταρχικός στόχος ε, η χρήση αυτή από πλευρά του Ταμείου. Θα έχω επαφή με τον συζητητή και τους σκιώδεις συζητητές για αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έληξε ο χρόνος στο Συμβούλιο. Θέλει να παρέμβει σύντομα στη συνέχεια των προηγούμενων παρουσιάσεων έτσι και στην πρόταση κανονισμού για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Αστυνομική Συνεργασία. Αύριο συνεδριάζει στο Συμβούλιο η Ομάδα Εργασίας για να ολοκληρωθεί και η τρίτη ανάγνωση με στόχο την επίτευξη μιας ικανοποιητικής και ποιοτική σύγκλησης σε επίπεδο του Συμβουλίου. Η Προεδρία χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής και της εισήγησης του κυρίου Γιακολίνο και ευχαριστεί επίσης την Επιτροπή για την προθυμία προς επίλυση και επεξήγηση των σημείων στα πλαίσια της σχετικής ομάδας εργασίας, όπως πράτηκε για τις υπόλοιπες προτάσεις των κανονισμών. Βέβαια, προς ενημέρωση μόνο ότι η πρόταση κανονισμού στο Συμβούλιο παρουσιάζει μια σημαντική εξέλιξη σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Οπότε και η παρέμβαση του κυρίου Γιακολίνο υπάρχει μια ε, ένα χάσμα σε σχέση με την εξέλιξη που βρίσκεται το κείμενο αυτή τη στιγμή βέβαια στο Συμβούλιο. Αυτό. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you, the presidency, Mr. Tavares. We're out of range in every possible way. The clock indicates... Κύριε Ταβάρες, ε, έχουμε περάσει το χρόνο μας. Θα θα είμαι πολύ σύντομος, ε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή Σαλβατόρο Γιακολίνο <clears throat> για ε, καλή σχέση σε σχέση με αυτή τη δουλειά που είχαμε. Αυτή δεν είναι απλή ε, έκθεση, είναι πολύ σύνθετη και περίπλοκη έκθεση. Είναι μια έκθεση που δεν μπορεί να εξεταστεί αποσυνδεδεμένα από τα διάφορα θέματα που αφορούν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε σχέση με την νομική βάση για τον χώρο Σέγγεν. Και θα ήθελα να καταστεί αυτό σαφέσα για όλους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό και υπάρχουν διάφορες διεκδικήσεις και αιτήματα σε σχέση με διάφορες εκθέσεις που έχουμε από πλευράς μας και σε σχέση με την Επιτροπή. Θα αναφερθώ σε σχέση με το θέμα αυτό και θα κατατεθούν τροπολογίες ώστε να μπορέσουμε να παρέμβουμε κατά το μέγιστο και αποτελεσματικά σε σχέση με αυτήν την έκθεση. Ένα στοιχείο θα ήθελα μόνο να σχολιάσω και αυτό είναι μεταξύ των διαφορετικών κριτηρίων που υπάρχουν και που καθορίζουν την ε, ουσία σε σχέση με τις δράσεις των ε, κρατών μελών και των κριτηρίων που αναφέρονται στο ΑΕΠ, ακαθάριστο εθνικό εγχώριο προϊόν, ή εγχώριο προϊόν κάθε χώρας και σε σχέση με την παρουσία ή όχι κρίσιμων υποδομών κέρια σημασίας που αποτελούν μέρος των υποδομών της Ένωσης. Πέρα από όλα αυτά, ο εισηγητής συμπεριέλαβε επίσης και τον διαχωρισμό των εσωτερικών συνόρων. Νομίζω θα άξιζε να σκεφτούμε καλά για τη συμπερίληψη αυτή ή όχι. Γιατί μπορεί να υπάρχει η ιδέα ότι κάποιοι υποφελούνται περισσότερο σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη και δεν θα θέλαμε να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό σε σχέση μέσα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο για μια πρώτη ανάγνωση, πρώτη προσέγγιση αυτού του εγγράφου που είναι κάτι που πραγματικά ε, έτυχε της προσοχής μου με μια πρώτη βιαστική ανάγνωση. Το Σεπτέμβριο σίγουρα θα υπάρξουν ευκαιρίες για να αναπτύξουμε περαιτέρω τη συνεργασία, το έργο αυτό με τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία που είχαμε και πιστεύω και ελπίζω ότι θα συνεχιστεί αυτή. Ευχαριστώ. Ε, σύντομα μπορείτε να αγνεύσετε καταφατικά, τίποτα άλλο, δεν χρειάζεται. Θα είμαι λακωνικότατος. Δύο σύντομες παρατηρήσεις για την αντίδραση της Κομισιόν. Ναι, το 50%, 50%, μεταξύ κρατών μελών και Κομισιόν. Υποθέτω ότι αυτό σημαίνει πως έχει οριμάσει η γνώση των κρατών μελών. Ε, θα πρέπει να τα ενθαρρύνουμε στα κράτη-μέλη για να χρησιμοποιήσουν ακόμα καλύτερα τους πόρους, ούτως ώστε αυτά πρώτα και καλύτερα να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις κρίσεις, να τις διαχειρίζονται καλύτερα. Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια, διάβασα το δελτίο υπαριθμών 2, ε, στο οποίο αναφέρθηκε η Κομισιόν. Παρακαλούμε την Κομισιόν να διαβάσετε και τους λόγους ε, που μας όθησαν να κατανείμουμε διαφορετικά τα κριτήρια. Ούτω ώστε και να λάβουμε υπόψη μας και τις μεταναστευτικές πιέσεις. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ένα ειδικό μέσο ειδικό για αυτές τις κρίσεις που αφορούν τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, αλλά μην ξεχνάτε πολύ συχνά οι μεταναστευτικές ροές είναι στα χέρια της μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό είναι λοιπόν το μέσο στο οποίο θα πρέπει να αναφερθούμε. Άκουσα τον κύριο Ταβάρες. Είμαι στη διάθεσή σας για απόλυτη συνεργασία να βρούμε την καταλληλότερη λύση, ούτως ώστε το κείμενο να γίνει συνεπές, ε, να λάβει υπόψη τις ανάγκες των πολιτών για την ασφάλεια που επιθυμούν και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Και κυρίως για τον, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κρίσεων. Σας ευχαριστούμε και εμείς κύριε Γιακολίνα για τη δουλειά σας και θα υποφεληθούμε από αυτή τη διαθεσιμότητα που δείχνετε για να συνεχίσει την εργασία, για να ολοκληρωθεί αυτή η έκθεση. Τώρα, οι προθεσμίες για τις τροπολογίες έχουν ε, καθοριστεί. Είναι η 5η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 12 καιρό το μεσημέρι. 5 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 12 καιρό το μεσημέρι. Σας υπενθυμίσω ότι ήταν πολύ εξαντλητική σημερινή μέρα. Δουλέψαμε πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποιες εργάσιμες την επόμενη εβδομάδα. Αλλά η, η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ συνεδριάζει σήμερα για τελευταία φορά πριν από τι καλοκαιρινέ διακοπέ. Θα ξαναρχίσουμε αρχέ Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα να σε ευχηθώ λοιπόν. Ο Αύγουστο. Να ξανα... Στον... Το Αύγουστο να είναι μια καλή ευκαιρία για να ξαναφορτώσετε τι μπαταρίε. Και να ξεχάσετε την εξαντλητική ψηφοφορία που χρειάστηκε να υποστούμε στην αρχή του απογεύματο. Πολλέ ευχές θα ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας αρχές Σεπτεμβρίου. Γεια σας.